Περίμενα μέχρι να έχουμε αρκετούς εισηγητές και σκιώδεις. Μου λέγουν ότι η μιλάει για το Σαΐρ και ο Διόγκο είναι εδώ. Φιλίπ, εσύ ο Σβέν. Είχα το θέμα του έστω. Α, ο Φιλίπ μάλιστα δεν μπορούμε να θυμόμαστε ποιος είναι ποιος εδώ πέρα. Καλωσορίζουμε τους πάντες. Είμαστε στο σημείο 6. Ετήσια έκθεση για τους φόρους. Όλοι Σμιτ, ενό συντάκτη του κειμένου. Συζητούμε τις τροπολογίες και θα δώσω το λόγο στον Όλε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης. Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ελπίζω ότι καταλήξαμε σε κάποιες επικοδομητικέ συμβαστικές λύσεις και ψηφίζουμε το απόγευμα, όπως γνωρίζετε. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα για να καλύψω σχεδόν όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι τις έχω καλύψει όλες στις συμβαστικέ όχι βέβαια τους πάντες σε κάθε συμβιβασμό, αλλά κάποιους τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά δίνει ένα μήνυμα ότι η πρώτη αυτή ετήσια έκθεση θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο βήμα να εξετάσουμε τις διάφορες ευαισθησίες. Είναι πολύ ευαίσθητα τα διάφορα ζητήματα, παρόλο που κατά διάρκεια των εργασιών είδα ότι πολλά από αυτά που συζητούσαμε ε, λίγο πολύ συζητήθηκαν σε άλλα βήματα συζητήσεων. Η φορολόγηση δεν είναι μόνο εσωτερικό θέμα, αλλά και ευρωπαϊκό. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και ίσως να καταλήξουμε σε κάποια άλλα συμπεράσματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλά. Εξετάσαμε σε ένα εργαστήριο τη διπλή φορολόγηση. Χρησιμότατο αυτό. Παρόλο που δεν μπορούσατε ίσως να συμμετάσχετε, θα έλεγα ότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε και να δείτε τις συζητήσεις. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες που ακούστηκαν. Δηλαδή ότι έπρεπε να υποστηρίξουμε την κινητικότητα κανονικά στην Ευρώπη και πολλοί φορολογούνται διπλά στην Ευρώπη. Υπήρχε κάποιος οδηγός φορτηγού στη Γερμανία. Εργαζόταν για τελική εταιρεία και δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα. Και όλο και περισσότερε τέτοιε διαμαρτυρίες, ε, καταγγελίες καταφθάνουν στην Επιτροπή Αναφορών. Πρέπει να το προσέξουμε. Δεν είναι μόνο θέμα που αφορά του συνταξιούχους. Αυτό είναι γνωστό θέμα, αλλά είναι ε, θέμα φορολόγησης και δεν είναι πρόβλημα μεθοριακό μόνο. Ε, δεν αφορά εκείνους που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές και ζουν σε μια χώρα και εργάζονται σε άλλη. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα πρέπει κάτι να κάνουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το έχει καταλάβει. Κάποια σχόλια για τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω να τις έχετε λάβει. Μάλιστα. Στην πρώτη συμβαστική για τις τηλογικές σκέψεις, την 1α, συμβαστική 1α, Συμπεριέλαβα την τροπολογία 12 του Καντράουι για τη σημασία που έχει το κράτο προνοία ε, τώρα τι εποχέ τη χρηματοπιστωτική κρίση. Στη δεύτερη συμβαστική για τι αιτιολογικέ σκέψει, αιτιολογική σκέψη 1 μάλλον, συμπεριέλαβα του, την τροπολογία 15 Γιώργη Κλούτε για την αποτελεσματική, την πραγματική φορολόγηση που είναι κάτι σημαντικό ε, για τις δημόσιες αρχές και την τοπολογία 16 του ΕΚΟΦΙΕΓΟ για τη σημασία για οι χώρες με ψηλό έλλειμμα ε, που έχουν, πρέπει να αυξήσουν τους, α, ε, τους φόρους που δεν βλάπτουν την ανάπτυξη. Στην τρίτη τη σημαστική 2, συμπεριέλαβα ε, τον Ήλκο κάπετ και την 17, 18 και 19 για κάποια ε, φορολογική ενοποίηση με κάποια θεμητή δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους ούτως ώστε να υπάρχει μια οικονομική εξοπιστία. Για τις παραγράφους συμβαστική 3α εκεί συνεργάζω του Γιώργ και του Φιλίπ της τροπολογία 29 και τη δική μου την επαριθμό 45 και προσπαθώ να περιγράψω το βασικό, τον πυρήνα του πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα. Συμβαστική 4 ε, ε, περιέλαβα τις τροπολογίες του Ραμών, του φίλου μου του φιλελεύθερου τη Βαρκελόνη και πρόσθεσα το ότι η φορολόγηση είναι κάτι που δεν αφορά μόνο την εθνική κυριαρχία αλλά μπορεί να είναι και θέμα περιφερειακής και τοπικής κυριαρχίας. Συμβαστική 5 συμπεριέλαβα κάποια τμήματα της τροπολογίας 41 του Σαΐτ και του Διέγκο την τροπολογία 36. Στη συμβαστική 6 συμπέλαβα την τροπολογία 52 και την 54, 53, την 55, την 56, την 57, την 58 και την 59 και νομίζω ότι είναι σημαντικό για χώρες με ελλείμματα να αυξήσουν τους φόρους τους ε, με έναν αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο και να επιδιώξουν ε, μείωση αποτελεσματική των δαπανών. Θα προτείνω σήμερα το απόγευμα και προφορική τροπολογία επί τη βάση της τροπολογίας του Diego την υπαριθμόν 64. Σημειώνω την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της φορολόγησης ε, για το FTB, για την βάση φορολόγησης και λοιπά και τον ενεργειακό φόρο και ήθελα αυτά ε, να αφήσω τη συζήτηση εκτός αυτής της οδηγίας. Η συμβαστική 6α ασχολείται με τη διπλή φορολόγηση, απάτε φορολόγηση και τη φοροδιαφυγή την 68 και την 69 συμπεριέλαβα του κυρίου Έπινγκ και, και το Ήλιο Κάλπελτ επίσης ε, υποστηρίζω την τροπολογία του έντρα Κιλούνα υπαριθμών 20 για τη σημασία που έχει η μείωση του κόστου συμμόρφωσης ε, προς τη φορολόγηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλωσόρισε και προς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εισαχθεί ε, ε θελοντικό CTB και την τροπολογία μου 72 και 73 που είναι τμήμα αυτής της συμβαστικής 7 μαζί με την τροπολογία 70 του Edward Σκυλούνα. Συμπεραίνει η έκθεση που πρέπει να βάλει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη για, πρασ, για το πρασίνισμα και το φόρο κατανάλωσης, από α, α, φορο, για τη φοροδιαφυγή, διπλή φορολόγηση ε, είναι στη συμβαστική παριθμών 8. Συμβαστική 9 Υποστηρίζω τις βελτιώσεις που προτείνει ο κύριος Έπινγκ και η κυρία Γκάλπελτ και ο κύριος Φέγιο, την 102 δηλαδή. Θα έχουμε και άλλη προφορική τροπολογία του Ντιέγκο για τη διπλή φορολόγηση, τροπολογία 107. Ε, είναι σημαντικό οι πληροφορίες που παρέχονται στους πολίτες να είναι γραπτές σε φιλικές προς το χρήστη μορφή και συμβαστική 10 έχουμε το κείμενο του κυρίου Έπιν και του κυρίου Φέγιο. Συμπεριλαμβάνονται τα κείμενά τους. Κάνω ό,τι μπορώ, βλέπετε. Υποστηρίζω τμήματα της τροπολογίας της Άλλη Μακάρθη, της 136, για τη σημασία που έχει κατά πολέμηση της φοροαποφυγής και θα υποβάλουμε σχετικώ προφορική τροπολογία αν κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό. Το κάτω μέλο θα πρέπει να δράσει στη 11 11β και τέλος θα πρέπει η οδηγία να ολοκληρωθεί για την εξοικονόμηση από το φορολόγηση και να υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Υποστηρίζω λοιπόν την 144, την τροπολογία του Φιλίπ που αναφέρεται στο θέμα. Υποστηρίζω και μέρη τη δική του τροπολογία Φιλίπ στην 153 και προτείνω προφορική τροπολογία που σχολιάζει το τελευταίο κομμάτι αυτή. Ένα από τα δυσκολότερα, οι συμβιβασμό αφορούσε του φορολογικού παραδείσου αλλά ελπίζω ότι θα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Καλούμε τα κάτι μέλη να δώσουν ύψη στην προτεραιότητα στο θέμα. Ξέρω ότι αυτό είναι ευαίσθητο ε, ζήτημα. Συμβαστική 11α όσον αφορά του φορολογικού παραδείσου, τροπολογία 83, 138, 155 και 156 ε, λαμβάνονται υπόψη και κάποια σχόλια που αφορούν τι μεμονωμένε τροπολογίε που δεν συμπεριλαμβάνονται στι συμβαστικέ τροπολογίε. Όπω προανέφερα, δεν είμαι υπέρ τη τροπολογία που καλύφθηκε το FTT και το ΦΠΑ λεπτομερώ. Ε, ε, και το φόρο δηλαδή των χρηματοστοτικών συναλλαγών καλύπτονται αλλού. Έχουμε και την έκθεση τη Άννα Ισποδηματά όσον αφορά το, τη φορολόγηση των χρηματοστοτικών συναλλαγών. Άρα δεν υποστηρίζω τι σχετικέ τροπολογίε που υπευλήθησαν. Ε, υπάρχουν αρκετές από αυτές που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα και θα τις δείτε. Είναι πιο ρεαλιστική η προσέγγιση που ακολουθούμε τελικά. Αναγνωρίζω ότι ο οικονομικός φεντεραλισμός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και φορολογικός φεντεραλισμός και έχω να προτείνω φορολογική τροπολογία Ο Ραμόν δεν είναι εδώ. Αλλά ίσω κάποιος από ομοσπονδο, ομοσπονδιακό κράτο θα πρέπει να μα πει πως βλέπουν το φορολογικό φεντεραλισμό ε, διότι και αυτό είναι ευαίσθητο θέμα είναι ευαίσθητη διατύπωση έκφραση τι σημαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μου έχουμε τοπικό φόρο και περιφερειακό φόρο, αλλά συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο και διανέμονται προς την τοπική αυτοδίκηση. Τέλος, ελπίζω ότι αυτή η πρώτη ε, έκθεση για τη φορολόγηση του Κοινοβουλίου θα πιέσει κάπως τα κράτη-μέλη, ούτε ώστε να υιοθετήσουν τάχιστα τις υφιστάμενες προτάσεις για τη φορολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω και αυτό είναι μέρημνά μου ότι αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποβάλει σχετικέ προτάσει για την λύση συγκεκριμένων προβλημάτων που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτε και οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινά. Οπότε θα ήθελα να κλείσω εδώ και για μία ακόμη φορά θα ήθελα να εκφράσω την, ε, τις μου προς τους κοιόδης εισηγητές και τους βοηθούς τους ε, διότι νομίζω ότι πρέπει να πω δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα και ελπίζω ότι στο τέλος ε, θα καταλήξουμε σε ένα λογικό ανεκτό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ωραία, λέει η πρόεδρος. Ο Διόγκο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας τον ε, Όλε και να τον ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για αυτό το πεπλεγμένο θέμα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις που ήταν δύσκολες σε πολιτικό επίπεδο ακόμα και μέσα στις ίδιες πολιτικές ομάδες είχαν αφιλεγόμενο χαρακτήρα τον ευχαριστώ λοιπόν για την πάρα πολύ σημαντική εργασία που έχει κάνει σαν εισηγητή, για το γεγονό ότι έμεινε πάντα σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές και για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Στην πρώτη τώρα αυτή έκθεση που αφορά τη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να έχει μια θετική, μια σημαντική έγκριση στην ψηφοφορία του απογεύματος και γι' αυτό θέλω να εξάρω τις προσπάθειες που έχουν γίνει από όλους αυτούς που συμμετέσχαν σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές η επαφή μας έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω προτάσεων που ήταν καινοτόμε και ήρθαν τελευταία στιγμή, αλλά χάρη στις ε, τεχνολογίες της πληροφορίας όλοι είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε κοινωνοί του και να δώσουμε την αντίδρασή μας. Για τα θέματα τώρα αυτά της φορολογίας. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο συλλέγει ομοφωνία μέσα στο κοινοβούλιο μας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Πολλές φορές αυτό προκύπτει και από την προέλευση των βουλευτών και φυσικά και από την κατάσταση οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε και τίθεται το ερώτημα ποιος πρέπει να είναι μέσα στην κρίση αυτή ο ρόλος της φορολογίας σε χώρες που έχουν μεγάλο εξωτερικό, μεγάλο χρέος, σε χώρες που έχουν μεγάλο έλλειμμα. Τι ρόλο λοιπόν μπορεί να παίξει η πολιτική φορολόγηση <clears throat> για να αντιμετωπίσει την κρίση και να μας βοηθήσει να εξέλθουμε από την κρίση. Υπάρχουν οι απόψεις ιδιαίτερα φιλελεύθερες και οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει ε, μια σειρά θυσιών των πολιτών μέσω της φορολογίας. Και αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πέραν αυτού του γενικού θέματος, του ρόλου της φορολογίας, Υπήρξε και ένα άλλο πλέγμα θεμάτων τα οποία συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής της έκθεσης. Αντιμετώπιση της απάτης και της ε, φοροδιαφυγής. Το θέμα του δημοσιονομικού φεδεραλισμού. Αυτή είναι μια έννοια την οποία χρησιμοποίησαμε εμείς για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή έννοια Δεδομένου ότι έχουμε μεγάλες διαφορές μέσα στα κράτη-μέλη. Στην Πορτογαλία όλοι οι φόροι αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους φόρους ε, συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για φόρους που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς δήμους και κοινότητες. Έχουμε λοιπόν φόρους σε επίπεδο κρατικό και φόρους σε επίπεδο τοπικό, δημοτικό, αλλά είναι διαφορετική κατάσταση σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αντίθετα από άλλες χώρες, στην Πορτογαλία όλοι οι φόροι συλλέγονται σε κεντρικό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης και άλλες προκλήσεις <clears throat> οι οποίες αναδύονται και ένα τμήμα της εργασίας μας ήταν να καταγράψουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Μιλάμε πάρα πολύ για θέματα προσωπικής φορολογίας, φορολογίας προσωπικού εισοδήματος ή φορολογίας κατανάλ, της κατανάλωσης όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή φορολογία. Αλλά υπάρχει και το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων. Πώς θα φορολογηθούν επιχειρήσεις που έχουν θηγατρικές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι πάντα στην ίδια χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε καλύτερα για το μέλλον και υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Συνολικά λοιπόν αυτή η έκθεση θέτει ανακλήφω όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανταλλαγή πληροφοριών, το ΦΠΑ, και στη συνέχεια <clears throat> ξεκινάει <clears throat> τη συζήτηση για τις μελλοντικέ προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γνωρίζοντας ότι μέσα σε αυτά τα θέματα, την αντιμετώπιση των προκλήσεων, υπάρχουν βαθιές ιδεολογικές διαφορές και επίσης διαφορές που οφείλονται στη γεωγραφική προέλευση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έργο μας λοιπόν το πολιτικό είναι ένα πάρα πολύ θετικό έργο γιατί εστιάζεται στο κοινό πυρήνα που έχουμε όλοι ως Ευρωπαίοι για αυτό το θέμα της φορολογίας που είναι τόσο σημαντικό και θέλω να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρος. Η, η Ανακάρτη. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΑΙΝΤ, ο οποίος είναι ο συντονιστής στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου ψηφίζουν αυτή τη στιγμή. Θα διαβάσω λοιπόν τη δήλωσή του. Σας ευχαριστώ πολύ, τον, ε, ιδιαίτερα τον εισηγητή, και για τις ε, συμβαστικές λύσεις που επετέθησαν. Θεωρούμε τα κύρια προβλήματά μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους φορολογικούς φραγμούς, τη φοροδιαφυγή και να έχουμε νέους ε, βιώσιμους πόρους. Είναι σημαντικά τα σχόλια του κ. Σμιτ και λαμβάνει υπόψη πολλές από τις απόψεις μας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι συμβαστικές λύσεις απαιτούν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τους φορολογικούς παραδείσους και όχι μια συμφωνία σε επίπεδο κρατών μιλών. Επίσης χαιρόμαστε για την ιδέα του να υπάρξει σαφή προσδιορισμό του τι σημαίνει φορολογικός παράδεισος και επίσης να εξασφαλιστεί μια πιο αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα φορολογικά ζητήματα. Θα θέλαμε επίσης να έχουμε δει στην έκθεση μια πιο στεναρή δήλωση για την ανάγκη να υπάρχει μια πιο ε, σημαντική συμμετοχή του six του ε, εξαμερούς ε, νομοθετήματο στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να δώσουμε ένα πιο ενεργό ρόλο στη Eurostat για τη συλλογή φορολογικών δεδομένων και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση της Επιτροπής μας και του Ευρωκοινοβουλίου για τη φορολογική πολιτική. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που την ανέλαβε ο Όλη Σμιτ. Όλοι νομίζω ότι μπόρεσες να περάσεις στην ουσία του θέματος, θέτοντας τα θεμέλια της πραγματικής δουλειάς που πρέπει να γίνει για τους φόρους. Το πραγματικό ζήτημα λοιπόν είναι αν θα έπρεπε να συμφωνήσουμε ή όχι και αν μπορούμε σε κάποιες βασικές αρχές για τη φορολογία. Λόγω χάρη είμαστε κατά τη διπλή φορολόγηση, αλλά εξίσου και κατά τη ε, απάτης ή της προδιαφυγή. Αυτά όλα είναι πολύ ξεκάθαρα χάρη στην έκθεση που συνέταξε. Και έδωσες, ε, προσέφερες τη βάση για μια συμφωνία ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον βάσει των συνθήκων ή θεωρητικά δεν έχουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στο θέμα αυτό. Άρα ο μόνος τρόπος να βαρύνει η απόψή μας ήταν να μιλήσουμε με νέα φωνή. Θα στηρίξουμε λοιπόν την έκθεση και τις συμβαστικές προτάσεις. Απλώς μια μικρή λεπτομέρεια σε μια αιτιολογική σκέψη. Όταν στην αιτιολογική σκέψη ή στην ε, συμβαστική σου ένα α μιλάμε για περιβολικό χρέο των κρατών μελών. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά, Ακούμε ότι μόνο, το μόνο αίτιο για την ε, σημερινή κρίση είναι τα κρατικά χρέη. Θα προτιμούσαμε να αναφέρετε λοιπόν και το κρατικό και το ιδιωτικό χρέος και οι οικονομικές ε, ανισορροπίες οι οποίες έχουν να κάνουν βέβαια με το κρατικό χρέος αλλά και το ιδιωτικό αλλά και η έλλειψη ισορροπίας στην ανταγωνιστικότητα και το καθεξής. Για μένα είναι πολλαπλές οι αιτίες της κρίσης. Τώρα ως ομάδα Δεν μα πειράζει να μην αναφέρονται όλα τα ζητήματα περί φορολογικής πολιτικής, διότι από τη μια δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το six-pack, αλλά δεν ανάγκη να το παραλαμβάνουμε σε κάθε μια έκθεση που γράφεται από εδώ και στο εξή. Δεν με πειράζει λοιπόν να με αναφερθεί και εδώ. Τελευταία παρατήρηση για το φορολογικό φεντεραλισμό. Καλά κάνεις και το αναπτύσσεις, όμως είναι τρίπτυχη νομίζω αυτή η έννοια. Πρώτον, λέει ότι ως τώρα είχαμε τρία επίπεδα για τη φορολογία, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν τέσσερα. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κάποιο, απλώς θέλουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο να προσθεθεί στα προηγούμενα. Και εκεί μπορεί να έχει νόημα να επιβληθούν φόροι. Έπειτα, χρειαζόμαστε δύο στοιχεία σε ένα πραγματικό φορολογικό φεντεραλισμό. Πρώτα απ' όλα κοινού κανόνες και αυτό σημαίνει κανόνε για τη φορολογική βάση και τα, τους και έπειτα ε, περιθώρια λιγμού σε κάθε επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή θα έχουμε ένα ενιαίο μοντέλο για όλα τα επίπεδα. Θα υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, αλλά ευέλικτο. Δεν θα μπορούμε να είμαστε αδιάλεκτοι και όλοι να επιβάλλεται να κάνουν τα ίδια. Και έπειτα στην φάση της συλλογή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη η διοίκηση οργανώνεται σε επίπεδο κράτους μέλους για τη συλλογή των φόρων. Ίσως πρέπει κάτι νέο να επινοήσουμε. Η συλλογή καλώς θα πρέπει να γίνεται και στο μέλλον στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά ίσως η διανομή να μην γίνεται μόνο προς το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και προς το ομοσπονδιακό εφόσον χρειαστεί. Εάν λόγου χάρη αποφασίσουμε ότι θα υπάρξει ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή κάτι άλλο που θα επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τέλο πάντων για τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της φορολόγησης εφόσον αποφασιστεί. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν ξανά για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξες. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που αρέσει ο διάλογος και για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ για τη δουλειά που έκανε. Δεν είναι εύκολο να συμφιλιώσει κανεί τι ε, πολύ διαφορετικέ απόψει που υπάρχουν στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη φορολόγηση. Και σήμερα υπογράμμισα, ε, τις, ε, υπογράμμισε μάλλον τις, ε, τις τροπολογίες που υποστηρίξει η ECR. Τροπολογία 1 και 2 για, για την πραγματική φορολόγηση και την δημοσιονομική ενοποίηση ε, είναι τη λογική σκέψη που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Θα υποστηρίξουμε και συμβαστικέ τροπολογίε 3, 6α και 11 για τι φορολογικέ πολιτικέ κατά τη διπλή φορολόγηση, φορολογικών απατών και φοροδιαφυγή για να βρεθούν λύσει για αυτά τα προβλήματα και να μειωθούν οι διοικητικέ αβεβαιότητε για τι επιχειρήσει και του πολίτε και χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτω μελών. Τρίτον, συμβαστικέ 9 και 10 είναι ιδιαίτερο σημαντικέ διότι εστιάζονται επί τι εμπειρίε των πολιτών με τι εφορίε, με τι φορολογικέ αρχέ ερωτηματικά που έχουν οι πολίτε με θέματα που αφορούν τους φόρους που θα πρέπει να απαντώνται εγκαίρω από τι αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να καλύπτεται μέσω ε, μιας ε, ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ενώσεω όπου θα μπορούν οι χρήστε να βρουν σε φιλική μορφή τι πληροφορίε που χρειάζονται όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές ε, και τι διάφορε πληροφορίε για του φόρους. Μετά έχουμε άλλε τρει σημαντικέ λύσει που θα υποστηρίζαμε εάν είχαν αλλάξει κάποια μικρά τμήματα, όπως συμβαστική 4, όπου δεν επιτρέπει δημοκρατικό έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια τώρα. Επιπλέον δεν συμφωνούμε με την αρμόνιση των φόρων που θεωρείται σε βασικός παράγον για την ανάπτυξη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη Συμβαστική 5. Ο κύριος Σμιτ και ο κύριος Κλίμς θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η αρμόνιση φορολογική οδηγεί σε υψηλότερη φορολόγηση και σκοτώνει τις δουλειές. Ο ανταγωνισμό ο φορολογικό που υποστηρίζω εγώ ε, πιέζει προ τα κάτω του φόρου και δημιουργεί θέσει απασχόληση. Άρα ε, είναι το αντίθετο το κείμενο από αυτό που θα είναι τα περισσότερα μέλη. Στο βασιστική 11β είμαστε υπέρ ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια τη οδηγίας για εξοικονομήσει όσον αφορά τους φόρους ε, αλλά αμφισβητώ κατά πόσο θα πρέπει να γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτόματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω άλλο να θέλει να μιλήσει, οπότε επιστρέφουμε σε σένα όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ τα σχόλιά σας και νομίζω ότι συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι συμφωνούμε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές βέβαια και θα υπάρχουν. Και εναλλακτικές. Πάντα είναι καλές οι εναλλακτικέ. Η διατύπωση όμως είναι το βασικό. Συμφωνώ με τον Φιλίπ. Εάν θέλουμε να έχουμε κάποια επιρροή, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια συνένεση εντός της Επιτροπής αυτής. Διότι αν μελετήσουμε κάθε κείμενο, κάθε τροπολογία, ακόμα και στην ομάδα των φιλελευθέρων, θα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Συνηθισμένο αυτό. Πραγματικά ελπίζω ότι θα πετύχουμε ευρεία συνένεση στο τέλος και θα εξετάσω την αιτιολογική σκέψη 1α και αυτός ο δημοσιονομικός φεντεραλισμός διερωτώ με αν ήταν το νόημα, το πνεύμα της πρότασης αν αυτό είναι το νόημα Ίσως τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Προσπάθησα, τουλάχιστον, με κάποιες μικροαλλαγές να δεχτώ τις τροπολογίες του Ραμών και άλλων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ψηφίζουμε το απόγευμα και στόχος μας είναι η Ολομέλεια η δεύτερη του Φεβρουαρίου Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά. Πάμε στο σημείο 7 αφορά τους οίκους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Ο, ο Λεωνάρδο λοιπόν, Ντομένιτσι είναι ο συντάξη του κειμένου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχω στη διαθεσή μου, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Α, το θέμα τον οίκων αξιολόγησης ε, παρουσιάζεται ιδιαίτερα περίπλοκο και ευαίσθητο. Είναι ένα ζήτημα άκρος επίκαιρο. Μίλησε χτες γι' αυτό και ο πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το ότι υπάρχει μεγάλη απέτηση ρυθμίσεως στον τομέα αποδεικνύεται και από τις διάφορες ε, διατάξεις που υποβάλλονται, ξεκινώντας από πρώτο κανονισμό του Νευρίου του 2009 από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στο δεύτερη, στην αναθεώρηση του Μαΐου 2011 μέχρι ε, τον τελευταίο κανονισμό που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος τον Νοέμβριο. Ε, υπενθυμίζω όλος ιδιαίτερος ε, τη δουλειά που έγινε από αυτών των ζητημάτων από τον συνάδελφο Γκοζές σε αυτή την Επιτροπή και φυσικά υπενθυμίζω και την έκθεση κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας που ετοίμασε ο συνάδελφος Βολφ Κλίντς. Σημερίζομαι συμμερίζομαι ε, τη γενική προσέγγιση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα υποστηρίζονται από τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Η προσέγγιση δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια ε, λογική ιδεολογική ούτε μια λογική επιβολής κυρώσεων. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πολυάριθμα σφάλματα που έχουν διαπραχθεί στις αξιολογήσεις από πλευρά των οίκων αξιολόγησης, rating κατά το παρελθόν, που προφανώς απαιτούν ε, κριτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους. Και αναφερόμενος ε, σε μία πιο πρόσφατη περίοδο, θα ήθελα να πω πρέπει να δούμε και το χρονισμό των αξιολογήσεων, κυρίως ε, όσον αφορά τα κρατικά χρέη, που πολύ συχνά υπονοούν και βλέπουμε να διαφαίνεται μία προσπάθεια επιρροής, επηρεασμού απαραδέκτου ε, όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται και σεισμικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι από αυτή την επόψη είναι σημαντικό η πολιτική και τα θεσμικά όργανα να αναλάβουν τον ε, ρόλο τους ε, και να κάνουν δύο ρυθμίσει. Τα βασικά στοιχεία της πρόσφατης προτάσεω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αφορούν την over-reliance, υπερβολική εξάρτηση ε, από τους οίκους αξιολόγησης και δεύτερον είναι κάτι που αφορά και το θέμα της αξιολογήσεως των κρατικών χρεών τη σύγκρουση συμφερόντων, την κυκλική εναλλαγή για την υποστήριξη του ανταγωνισμού, την απαγόρευση των, της αξιολόγησης επί εταιριών που, που, στις οποίες υπάρχει συμμετοχή, αστική ευθύνη, τη στιγμή κατά την οποία διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβιάσεις. Επί κάθε προναφερθέντος σημείου νομίζω ότι είναι τα τη ε, μια αντελεχής ανάλυση από πλευράς ε, της Επιτροπής μας και θα ήθελα να μπορέσω να βασιστώ στη συνεισφορά όλων των συναδέλφων ξεκινώντας από τους εισηγητές με τους οποίους με μερικούς από αυτούς τουλάχιστον ήδη είχα κάποιες ε, επαφές. Πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε κάποια σημεία και να εμβαθύνουμε σε αυτά με στόχο την βελτίωση της ε, λειτουργίας του οικονομικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο καθένας έχει τις ιδέες του πάνω σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι δυνατόν επ' αυτού να βρούμε μια κοινή βάση συνεννόησης. Διατηρώντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά συνεισφέροντας εμείς ως Κοινοβούλιο στην επεξεργασία νέων ιδεών και νέων προτάσεων και ε, ε, από τη στιγμή που είναι βέβαια είναι ξεκάθαρη στόχη, αλλά είναι λιγότερο ξεκάθαρο και πιο δύσκολο να βρεθεί τρόπος να μεταφραστούν σε νέους κανόνες αυτές οι αρχές και αυτή η στόχη, η γενική στόχη. Πιο συγκεκριμένα, εγώ τέσσερα σημεία που θα πετήσουν κατά την άποψή μου ε, μία εμβάθυνση ιδιαίτερη, συγκεκριμένη. Εμπρότης ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο που αφορά το κρατικό χρέος και τις σχετικές αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης για τα κρατικά χρέη. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη εισάγει κάποια στοιχεία καινοτόμα και σημαντικά όπως επί παραδείγματι το συχνό rating όσον αφορά τα κρατικά χρέη κάθε έξι μήνες και δώδεκα μήνες. Ε, την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες πληροφορίες επί των κριτηρίων που υιοθετούνται και μέσω της δημοσίευσης κριτηρίων που θεσπίζονται για αυτές τις αξιολογήσεις, τα ratings και τη δυνατότητα που προσφέρεται στα κράτη που υπόκεινται σε αξιολόγηση να εκφράσουν τις θέσεις τους πριν να ανακοινωθούν οι αξιολογήσεις αυτές καθ' Εγώ πεθυμίζω ότι επί του συγκεκριμένου ζητήματος ήδη διεξήχθη η συζήτηση εντός του σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο του κανονισμού αφαιρέθηκε η δυνατότητα να δίνεται εξουσία στην ΕΣΜΑ να αναστέλει την οικονομική αξιολόγηση των χωρών κατά την περίοδο κατά την οποία ε, έχουν, ε, εφαρμόζουν σχέδια εξυγίανσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε εις βάθος όχι για να το επαναπροτείνουμε έτσι μηχανικά στη συζήτησή μας ή στην πρόταση που θα υποβάλουμε τελική, αλλά διότι παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βρεθούν νέες λύσεις σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά τις χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και που τελικά αξιολογούνται, υπόκειται στο rating. Ε, άλλο σημείο ε, για το οποίο χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να γίνει δελεχή συζήτηση είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι εγώ είμαι υπέρ του πνεύματος που διαπνέει το κύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να ανοίξει η αγορά που ε, θα ελέγχεται κατά 90%, που ελέγχεται κατά 90 από τις τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης εγώ νομίζω ότι θα πρέπει προσεκτικά να αξιολογήσουμε τις συνέπειες του συστήματος της, το, της, της εναλλαγής που προτείνεται, της κυκλικής εναλλαγής. Δηλαδή κάθε τρία χρόνια εκ περιτροπής να εναλλάσσονται οι οίκοι οι οποίοι θα κάνουν την αξιολόγηση και επίσης και η περίοδος cooling off όπως αποκαλείται που ε, θα πρέπει να είναι τετραετής. Σαν τρίτο σημείο, όσον αφορά τη σύγκρουση των συμφερόντων, ε, πιστεύω ότι χρειάζεται από την πλευρά μας να εμβαθύνουμε στο θέμα των ενδεχομένων εναλλακτικών σε σχέση με το Issue Spain Model. Δηλαδή, να μπορούμε επί τη βάση διαφόρων πολλών προτάσεων μάλλον που έχουν υποβληθεί να αξιολογήσουμε το θέμα της χρήσεως μέσων που θα ε, ευνοούν ένα investors model. Τέταρτο σημείο ε, θα πρέπει ενδελεχέστατα να δούμε πώς μπορούμε προβούμε σε μία πλήρη αναθεώρηση του συστήματος κανόνων και νομοθεσιών που υπάρχουν που ευνοούν την υπερβολική εξάρτηση, το over-reliance και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην εναρμόνιση ε, των συστημάτων που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και κυρίως σε σχέση με την νέα νομοθεσία που λειτουργεί και εφαρμόζεται στις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα σημείο ιδιαίτερα περίπλοκο, κυρίως διότι έχει πολλές τεχνικές συνέπειες που πιστεύω ότι θα απαιτήσουν ιδιαίτερη εμβάθυνση. Και τέλος, μια τελική παρατήρηση πριν ολοκληρώσω. Ε, κατανοώ τις δυσκολίες σχετικά με την πρόταση να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή υπηρεσία αξιολόγησης, rating, και καταλαβαίνω και τους λόγους για τους οποίους δεν προωθείται αυτή η πρόταση στο νέο ε, κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η πρόταση. Όμως δεν θεωρώ θετικό το ότι δεν υπάρχει καν μία αναφορά στην προώθηση μίας ή περισσότερων οίκων αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κατά την άποψή μου παρά το περίπλοκο χαρακτήρα του θέματος θα αποτελούσε ένα σημαντικό στόχο προς επιδίωξη. Σταματώ εδώ για να αφήσω χρόνο στους συναδέλφους να συμβάλλουν στη συζήτηση. Το θέμα είναι περιπλοκότατο. Όπως προανέφερα, ελπίζω να μπορέσω να χρησιμοποιήσω, να εκμεταλλευτώ, να βοηθηθώ από τη συνεισφορά των συναδέλφων. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που προβλέπει μια κρόαση στις 24 Ιανουαρίου μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών για 22 Μαρτίου και μια ψήφος στην Επιτροπή στις 21 Μαΐου. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικός στόχος αυτός να καταφέρουμε να εγκρίνουμε το νέο κανονισμό μέχρι το καλοκαίρι. Ε, και υπογραμμίζω αυτό το θέμα διότι πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερά μας προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το πρόβλημα ε, των αργών ρυθμών των διαδικασιών λήψης αποφάσεω που μαστίζουν σε αυτή, σε αυτή τη φάση που φρενάρουν τις σημαντικές, ε, σημαντικούς νόμους που θα έπρεπε να θεσπίσουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Jean ευχαριστώ, Jean Πολ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καθησυχάσω καταρχήν τον εισηγητή, όπως είχαμε κάνει και προηγουμένως σε μια διμερή συνομιλία ότι θα τον βοηθήσω και ότι είμαι όπως και αυτός αποφασισμένος να εξασφαλίσω την αποτελεσματικότητα και τον παραγματιστικό χαρακτήρα κάθε στα θέματα αυτά. Θέλω όμως να σταθώ σε ορισμένε παρατηρήσεις οι οποίες δεν αντιφάσκουν με αυτά που λέει ο εισηγητής, πιστεύω ότι συμπληρώνουν τη σκέψη του. Ρεαλισμός καταρχήν. Είπατε προηγουμένως αγαπητέ φίλε ότι παρακολουθήσατε από κοντά τους δύο προηγούμενους κανονισμούς, αλλά θα ήθελα σήμερα να σας εξηγήσω πώς έτυχαν έγκρισης οι τρεις μεγάλες εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό θέμα, όπως βλέπετε. Δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, είναι πολύ πολιτικό. Ο πρώτος κανονισμός για τους 20 αξιολόγησης προέβλεπε μια έγκριση για ένα λειτουργήμα που μέχρι τότε δεν υφίστατο κανένα έλεγχο. Υπήρχε τότε η, η ΕΣΜΑ η αρχή των ε, ε, αγορών κινητών αξιών. Η ΕΣΜΑ λοιπόν μετά από την έκθεση Λαροζία δημιουργήθηκε, αλλά ο πρώτος της κανονισμός θεωρούσε ότι ήταν απλώς ένα σώμα ρυθμιστών και εποπτών που θα παρακολουθούσε όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθηθούν και να ελεγχθούν μέχρι ότου υπήρχε ένας αντίστοιχος φορέας ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τη σκητάλη. Τότε οι τρεις αυτοί φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης υπέβαλαν τα διαπιστευτήριά τους το Σεπτέμβριο του 2010. Τον Μάιο του 2011 δεν είχαν ακόμα τύχη έγκρισης. Έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της ΕΣΜΑ και στον επίτροπο κ. Μπαρνιέ να τονίσω ότι είναι παράξενο η μόνη αυτή ρύθμιση που έγινε μετά από την κρίση να μην εφαρμόζεται. Και μου <clears throat> απαντήσανε από τη μεριά του κ. Μαγιέρ ότι υπήρχε και ένας ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης ο οποίος επρόκειτο να εγκριθεί. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς είχε πει αυτός ο ιαπωνικός οίκος για το κρατικό χρέος. Πέρασε το καλοκαίρι του 2011, υπήρξαν συζητήσεις στην Ολομέλεια με παρουσία και του κυρίου Μπαρόσο, το είπα στον κύριο Τρισσέ στην τελευταία του παρουσία για τον νομισματικό διάλογο και εντυπωσιάστηκε που δεν είχε υπάρξει ακόμα αυτή η έγκριση των πιστοληπτικών οίκων. Το 18 Οκτωβρίου ο κύριος Μαγιέρ ήλθε να με επισκεφθεί και μου ζήτησε να σταματήσω τα πειρά εναντίον του γιατί <clears throat> θεώρησε ότι τον ενοχλούν αυτά τα οποία λέω για την ε, ΕΣΜΑ. Είπε ότι δεν είναι το έργο μου αυτά τα πράγματα. Μα του είπα κανονικά εσείς θα συντονίσετε όλα αυτά. Αυτό είναι το έργο σας. Του, το ρώτησα τον κύριο Μάγερ αν θα μπορούσε να μου δώσει την εγγύηση ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Μου είπε δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Παράξενο, πριν από 8, μετά από 8 μέρες, μετά από αυτή τη συζήτηση, υπήρξε η έγκριση αυτών των τρίκων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ρώτησε τον κύριο Μπαρνιέ γιατί έγινε αυτό. Λέει γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτέ που μα τι πάνε και όλο ζητάνε να υπάρξει μια ανακοίνωση από τη μεριά τη Κομισιόν. Και αν θέλετε να προχωρήσετε αυτή την νομοθεσία, ίσω πρέπει να συμπεριφέρεστε με διαφορετικό τρόπο. Σα τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πόσο μεγάλη αδράνεια υπάρχει, αδράνεια από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, που καθυστέρησαν ιδιαίτερα για να αναλάβουν το σύνολο των ευθυνών τους σε σχέση με την εποπτεία των ενεργειών τους. Επίσης υπήρξε μεγάλη αδράνεια από τις ρυθμιστικές αρχές και φυσικά και από τις πολιτικές αρχές, γιατί εδώ μιλάμε για ένα θέμα ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η τάση αυτή στην Κομισιόν να θεωρούμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα του ανταγωνισμού με τεχνάσματα νομικίστικα εναλλαγή των φορέων αυτών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Όταν έχουμε τρει εταιρείε μεταξύ των οποίων εναλλασσόμαστε, δεν πάμε πολύ μακριά. Αν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστου οίκου αξιολόγηση, χρειάζονται πόροι και αξιοπιστία για αυτού του φορεί τα κράτη τα οποία διαμαρτύρονται για τους οίκους αξιολόγησης είναι τα πρώτα τα οποία τους ζητούν να αξιολογήσουν τα δικά τους ομόλογα. Και δεν το συστάνε από εθνικούς φορείς, αλλά από τους μεγάλους πιστοληπτικούς φορείς. Γι' αυτό είναι πολιτική λοιπόν η συζήτηση. Ενώπιον αυτής της κατάστασης είδαμε μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν τις προηγούμενες μέρες να περάσει αυτό το σχέδιο νομοθετήματος από την Κομισιόν. Ο Μισελ Μπαρνιέ, τον οποίο σέβομαι και αγαπώ πολύ, έκανε ό,τι χρειαζόταν, έκανε όλες τις απαραίτητες πράξεις επικοινωνίας μέχρι την τελευταία στιγμή που η μεγάλη πιστοληπτική οίκη ήρθαν στις 12 παρα 5 να του υπενθυμίσουν ότι τα μέτρα αυτά τα οποία ήταν έτοιμος να πάρει δεν ήταν τα κατάλληλα. Λοιπόν, νομίζω ότι το γεγονός αυτό ότι ελήφθη αυτή η απόφαση της Κομισιόν δεν ήταν η καλύτερη γιατί ήδη δημιουργεί μια κακή εντύπωση στις αγορές. Εγώ πρότεινα μια λύση για να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά με τρόπο ο οποίος να είναι λιγότερο υποκείμενο σε επικρίσει σε τεχνικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά να πράξουμε. Συμφωνώ και με τον συγητή όταν λέει ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα της ε, αμοιβαία συμμετοχής σε αυτές τις εταιρείες και της σύγκρουσης συμφερόντων λόγω ε, κατοχής μετοχών αυτών οι οποίοι αξιολογούνται. Το 2009 είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, η κυρία Μπέρες είχε κάνει μια σειρά προτάσεων για το θέμα αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε στην κατάλληλη λύση. Αν τελικά δεν υπάρχει το σύστημα ότι αυτός ο οποίος εκδίδει ένα αξιόγραφο, αυτός πληρώνει τους οίκους αξιολόγησης, τι θα γινόταν αν πρέπει να πληρώνει ο, ο επενδυτής, να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί στο ίντερνετ, θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τελικά η δράση των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι μια οικονομική δραστηριότητα σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι ο στόχος μας να απαγορεύσουμε να υπάρχουν αξιολογήσεις. Όλοι μας αξιολογούμε. Και εγώ όταν μιλάω με αξιολογείται. Δεν υπάρχει λόγος να εμποδίσουμε να υπάρχουν τέτοιοι φορείς οι οποίοι παίζουν το ρόλο των αξιολογητών για το λογαριασμό των επενδυτών. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην είναι μόνο αυτές οι πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται και μετά την κρίση της Ελλάδος να ακούμε όλοι μηχανιστικά τι μας λένε οι φορείς πιστοληπτική αξιολόγηση. Πρέπει να μας δίνουν απλώς στοιχεία πληροφόρησης και είναι πολιτική συζήτηση. Τι κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνησίων μας. Επικρίνουν τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά το πρώτο πράγμα που λένε είναι θα χάσουμε το τριπλό α ή θα πάρουμε το ένα ή θα πάρουμε το άλλο. Όταν λοιπόν ο υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία και το ενό πρόεδρο Γαλλική Δημοκρατία λέει: Άμα χάσω το τριπλό Α, θα χάσω τι εκλογέ. Αυτό είναι ηλίθιο. Δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα γιατί μετά από λίγο που φαίνεται ότι θα χάσει το τριπλό Α, λέει και τι έγινε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα άμα χάσουμε το τριπλό Α. Λοιπόν, οι φορεί αυτοί πρέπει να έχουν κάποιο ρόλο, αλλά αυτό το ρόλο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο νυφάλια και αυτό είναι ο δύσκολο ρόλο που έχει ο εισηγητή να μπορέσει να καταλήξει σε πραγματιστικού και συγκεκριμένου και αποτελεσματικού κανόνε ώστε <clears throat> να μπορέσουμε τελικά να απεξαρτηθούμε από αυτούς τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ευχαριστώ, ο Βολφ Κλίντς. Ευχαριστώ, Sharon. Είναι γεγονός ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης τους τελευταίους μήνες έχουν δημιουργήσει πολύ ντόρο γύρω από το όνομά τους. Όπως είπε ο Jean-Pierre δεν είναι μονάχα ένα σύνολο από τεχνικά ερωτήματα αλλά και πολιτικά ερωτήματα που συνάπτονται με αυτούς τους οίκους αξιολόγησης. Εγώ νομίζω όμως πρέπει να δούμε πιο αντικειμενικά τη συζήτηση για τους οίκους αξιολόγησης γιατί τον προηγούμενο μήνα ίσως κάπου βγήκαμε από τις ράγες και αυτό μας εμποδίζει να έχουμε μια σωστή κριτική στάση για τους φορείς αυτούς. Δεν ε, πρέπει να πυροβολούμε τον ε, αγγελιοφόρο που φέρνει τα κακανέα. Δεν είναι αυτή που είναι υπεύθυνη πάντα για αυτό το θέμα. Έρχομαι σε αυτό το οποίο την ανακοίνωση του Επιτρόπου κ. Μπαρνιέ. Έρχεται σε εύστοχη χρονική στιγμή, αλλά έρχεται συγχρόνως σε μια στιγμή που δεν ξέρουμε καν ο ήδη υπάρχον κανονισμός πώς λειτουργεί. Είναι γεγονός ότι χρειάστηκε πολλή χρόνος για να φτάσουμε σε αυτό τον κανονισμό. Εγώ συμμεριζόμαι πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν από τον Επίτροπο Μπαρντιά και περιλαμβάνονται στην ε, πρότασή τους, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία διαφωνώ μαζί του. Ξέρουμε καταρχήν ότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν κάνει λάθη μέσα στα πλαίσια της διεθνούς χρηματοπιστωτικούς ε, ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και αυτό οφείλεται σε ορισμένε περιπτώσεις επίσης στο γεγονός ότι υπήρχαν και εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων. Είχαν ακόμα και το γεγονός ότι πολλές φορές προέταξαν το εμπορικό του συμφέρον έναντι της ανάγκης αντικειμενικότητας. <coughs> και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Ιδίως όταν μιλάμε για θέματα ανταγωνισμού. Μέχρι την στιγμή που υπήρξε η κατάρρευση της Lehman Brothers, ήταν η κερδοφορία αυτών των φορέων πιστοληπτική αξιολόγηση 55% στο τζίρο τους. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα άλλο οικονομικό κλάδο. Μετά από την κατάρρευση της Lehman ε, Brothers ήταν ακόμα 30-35%. Λοιπόν, περνούσαν πολύ καλά αυτοί οι φορείς. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν για το ρόλο των μετοχών. Ποιοι είναι οι μέτοχοι οι οποίοι κρύπτονται πίσω από τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι μέτοχοι εφόσον υπάρχει μία ε, διαφάνεια και εφόσον δεν είναι καθαρά μέτοχοι μονάχα μιας από αυτούς τους, ε, της εταιρείας πιστοληπτικής ε, αξιολόγησης. Και εδώ υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν να ξέρουμε ποιοι από αυτούς τους μετόχους έχουν συμμετοχή πάνω από 5%. Είναι λοιπόν να μην υπάρχει διασταυρούμενη συμμετοχή αυτών των ε, μετόχων σε παραπάνω από μία εταιρεία και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συγχώρευσης αυτών των φορέων. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο περιορισμένος ο κανονισμό τη Κομισιόν. Λέει μονάχα για τα επόμενα 10 χρόνια. Εγώ δεν βλέπω την ανάγκη να υπάρχει χρονικό περιορισμό. Όταν έχουμε ένα ολιγοπόλιο τριών οίκων αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει συγχώνευση ή συνέργεια μεταξύ του. Επίση, για τον τομέα των οίκων αξιολόγηση, εμεί έχουμε προσπαθήσει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είχε απλώς χαρακτήρα δηλωτικό. Δεν υπήρξε, όπως ξέρουμε, καμία αντίδραση στην δήλωση προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει σε αυτή την περίπτωση να αναλάβουμε εμείς μια συγκεκριμένη ε, να αναλάβουν οι φορείς αναξιολόγηση, μια συγκεκριμένη ευθύνη και αστική ευθύνη για το έργο τους. <clears throat> να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει προσφυγή εναντίον τους στα δικαστήρια ε, επί τη βάση της αστικής ευθύνης που επέχουν. Αυτό είναι δύσκολο για μένα. <clears throat> Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι αποδεικνύεται λανθασμένη η κρίση μιας ε, εταιρείας πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο δίνει λαβή σε μια αστική αγωγή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην θεωρούσε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προφητεύει τι θα γίνει πάντα. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στοιχείο αστικής ευθύνη. Από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος ηθελημένα και ενσυνείδητα δρά προς το συμφέρον κάποιων μετόχων και κάνει χοντρά λάθη τα οποία δεν είναι απλώς τεχνικά σφάλματα αλλά είναι ε, ουσιαστικά σφάλματα. Δεν μιλάω για, την, ε, για το τεχνικό σφάλμα της υποβάθμισης της Γαλλίας που έγινε στο παρελθόν. Αν δεν υπάρχει λοιπόν καμία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν σωστά την αξιολόγηση, τότε μπορεί κανείς να μιλά για αστική ευθύνη αυτών των φορέων αξιολόγησης. Νομίζω το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι ελέγχουν το 95% της διεθνούς αγοράς. Υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις αξιολόγηση, αλλά οι τρεις αυτές είναι αυτές που κυριαρχούν στη διεθνή αγορά. Αν δούμε λοιπόν το θέμα από αυτή την οπτική γωνία, είναι γεγονός ότι η υπερβολική αυτή εξάρτηση από τους οίκους αξιολόγηση θα πρέπει να μειωθεί. Και εμείς έχουμε αυτό το καθήκον σαν νομοθέτες, γιατί έχουμε σε κανονισμούς καταγράψει ότι οι τράπεζες οι ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. θα πρέπει να επενδύουν μονάχα αν υπάρχει μια αξιολόγηση διπλό α ή διπλό α συν κτλ. Ενώ συγχρόνως λέμε στους κανονισμούς μας για τις τρεις αυτές συγκεκριμένες εταιρείες αξιολόγησης. Δεν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μία αξιολόγηση. Όχι, λέμε μία αξιολόγηση τη Moody's ή τη Standard Poor's ή τη Fitch. Λοιπόν, μετά δεν πρέπει να παραξενευόμαστε που οι εταιρείε αυτέ πηγαίνουν πρίμα στι δουλειέ του. Επομένω, εναπόκειται σε εμά να καταλάβουμε και να πούμε γιατί δεν έχουμε μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση και γιατί δεν αποκλίνουμε από αυτή την περιοριστική στάση και ζητούμε από τους ίδιους τους επενδυτές να κάνουν τη δική τους κρίση, να αποφασίσουν οι ίδιοι για το αν οι αξιολογήσεις αυτές είναι σωστές ή όχι. Γιατί μπορούν πάντα οι επενδυτές να βασιστούν σε πληροφορίες που έρχονται από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν θέλουν να κρίνουν για την φερεγγιότητα μιας επένδυσης. Τα δομημένα τώρα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Πολλές φορές χρειάζονται ειδικέ γνώσεις στα θέματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε τουλάχιστον δύο υποχρεωτικά αξιολογήσει Για να φτάσουμε σε αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καλύτερη μεθοδολογία. Και εδώ ίσως θα είναι πιο δύσκολο να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις φορείς αξιολόγησης. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και στα άλλα νομοθετήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Ε, στο παρελθόν θεωρούσαμε τα κρατικά ομόλογα είχαν μηδενικό κίνδυνο και αυτό οδηγεί και πάλι σε προβλήματα όπως αυτά που είδαμε με την εξάρτηση από τους οίκους αξιολόγησης. Έχω δύο ε, παρατηρήσεις. Καταρχήν το θέμα της εναλλαγής μεταξύ των οίκων αξιολόγησης προσωπικά. Όπως και ο Ζαν Πολ, θεωρώ ότι δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα αυτή η πρόταση. Όταν έχουμε μόναχα τρεις φορείς, και χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση δύο φορείς αξιολόγηση και λέμε ότι κάνουμε μία <clears throat> εναλλαγή, ουσιαστικά δεν αλλάζει αυτό ιδιαίτερο. Από δύο οίκου να περνάμε σε ένα παραπάνω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Επομένως αυτό δεν έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα η εναλλαγή. Αλλά θα πρέπει να δοκιμάσουμε αν θα μπορούσαμε αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο σε φορείς αξιολόγηση οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Αν θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν μονάχα οι τρεις αυτές μεγάλες εταιρείες αξιολόγηση, αλλά και άλλες οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ αποτελεσματικό ρόλο μέσα σε, στα κράτη-μέλη ή τις περιφέρειες των κράτους μέλους. Ε, και εδώ έρχομαι πάλι στο ρόλο της ΕΣΜΑ. Είναι σωστό να έχει τη δυνατότητα να κάνει αξιολογήσεις η ΕΣΜΑ, η Υπηρεσία Αγορών και Κινητών Αξιών. Αυτό είναι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδέα να προχωράει τόσο πολύ η εξέταση της ΕΣΜΑ, ώστε σε τελική ανάλυση να καταλήγουμε σε ταυτόσιμο μοντέλα από όλους. Δηλαδή δεν θέλω να ισοπεδώσουμε και να κάνουμε ταυτόσιμες τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από όλα τα πιστοτικά ιδρύματα και να έχουμε ένα ενιαίο μονάχα μοντέλο για την εκτίμηση της ε, αξιοπιστίας μιας επένδυσης. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 228 για τα κρατικά ομόλογα, το αν θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση μετά από 6 μήνε ή μετά από 12 μήνε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή πάντα οι οίκοι αξιολόγηση έρχονται κατόπιν εορτή και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Πώ μπορούμε να, να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι οι φορεί αξιολόγηση δεν χρειάζονται υπερβολικό χρόνο για μια αξιολόγηση αλλά μπορούν παράλληλα μέσα σε τρει-τέσσερι τρεις-τέσσερις ε, μήνες να κάνουν μια υποβάθμιση κατά τέσσερις ε, κλίμακες, τέσσερα σκαλιά της κλίμακας. Αυτά λοιπόν είναι τα κριτικά σημεία τα οποία ήθελα να θέσω και το ερώτημα, αυτό το οποίο λυπάμαι είναι το ερώτημα για το πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό το ερώτημα δεν εμφανίζεται καθόλου. Δεν θα μπορούμε να έχουμε αξιοπιστία χωρίς την επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού Πρέπει να μειώσουμε την πολιτική εξάρτηση. Δεν πρέπει να χάσουμε όμως την ευκαιρία να, κάνουμε μέτρα, να πάρουμε μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της αξιολόγησης και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απριόρι αδύνατο. Ε, Ευχαριστούμε. Ashley. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής να βελτιωθεί η διαφάνεια στον τομέα της αξιολόγησης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα και να υπάρξει περισσότερη δικαιοσύνη. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα δείκτη εδώ ευρωπαϊκή αξιολόγηση. η κεντρική συλλογή των πληροφοριών χρήσιμη θα ήταν, αλλά οποιαδήποτε τυποποίηση καταναγκαστική θα είναι ανταπαραγωγική προ τα μέτρα που θα στηρίξουν τον ανταγωνισμό. Όπω και ο κύριο Κλίντ, στηρίζω τα μέτρα για να μην υπάρχει υπερβολική εμπιστοσύνη στι αξιολογήσει. Θα πρέπει οι επενδυτέ να μπορούν να ασκήσουν τη δική του κρίση και όχι μόνο να επαφίονται στι τους οίκους αξιολόγησης. Πρέπει όμως να δούμε κατά πόσον θα κοιτάζουμε τι γίνεται με την εσωτερική αξιολόγηση για μικρές εταιρείε που ενδεχομένως να μην έχουν τέτοια εταιρική αξιολόγηση και τέτοιο σύστημα. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο μηχανισμός της υπερβολικής εξάρτησης από τις αξιολογήσεις ουσιαστικά αποσταθεροποιεί την αγορά. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να ενθαρρύνουμε την ε, συμμετοχή και νέων εταιριών, νεονίκων ε, αξιολόγηση επιστολητικής ικανότητας, αλλά όχι όχι ει βάρο τη ποιότητα. Συμφωνώ με τι παρατηρήσει Κοζέ και Κλίντ ότι δεν θα, αναγκαστικά δεν θα πετύχουμε καλύτερο ανταγωνισμό με τι περισσότερε εταιρείε. Θα πρέπει απλώ ε, μάλλον να περιμένουν ε, κάθε μια τη σειρά του για την επιρροή που θα έχουν. Εδώ λοιπόν η Επιτροπή θα πρέπει να ξαναδεί, σωστά έπρεπε να ξαναδούμε τι μεθοδολογίε ε, των οίκων που χρησιμοποιούν οίκοι αξιολόγηση και επίση να δούμε τι προτείνει και η ΕΣΜΑ για την τυποποίηση του συστήματο. Καλύτερο θα ήταν να υπήρχε μια ποικιλία μεθόδων. Το τελευταίο που θέλουμε είναι κάθε οίκο πιστολεπτική αξιολόγηση να ακολουθεί λίγο πολύ την ίδια μεθοδολογία. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα στρατιωτικά αποτελέσματα. Εδώ επίση να πούμε και για την ευθύνη των πολιτών Ίσως αυτό είναι μια από τις πιο βλεπερές συνέπειες της πρότασης, διότι είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και θέλουμε να υπάρξουν νέοι συμμετέχοντες στην αγορά, κυρίως μικρότεροι οίκοι, οι οποίοι να ανθίσουν. Εδώ λοιπόν, τι θα ήταν περισσότερο πετυχημένο, από το να επιβάλλουμε την κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη των πολιτών για όλους, την αστική ευθύνη για όλους τους ε, συμμετέχοντες. Αυτό μόνο θα έσπαγε την ε, καθεδρία των τριών. Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν εδώ σοβαρές βλαβερές συνέπειες. Η ασφάλεια για έναν μικρό συμμετέχοντα θα είναι σίγουρα ε, λιγότερο ανυπολόγιστες από αυτές για τους πάρα πολύ μικρούς. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι οπωσδήποτε να μην παραμείνει υπό το καθεδρία των τριών και να μην υπάρξει κατακαιρματισμός τη αγορά. Ο κ. Ντομινίτς βέβαια έχει δίκιο όταν λέει ότι οι οίκοι αξιολόγησεις έχουν κάνει μεγάλα ασφάλματα στο παρελθόν. Κυρίω για τα κρατικά χρέη. Ας θυμηθούμε όμως ότι αυτό που κάνουν οι εκεί είναι απλώ να γνωμοδοτούν. Δεν καταναγκάζουν κανένα να λάβουν υπόψη τις απόψεις τους, τις αξιολογήσεις τους. Ο λόγος που το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, οι επενδυτέ, είναι επειδή συνολικά συνήθως πέφτουν μέσα τις περισσότερες φορές. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ε, τα βάζουμε με τον αγγελιοφόρο των αυτών που μα δίνει απλώ πληροφορίε, Έχει βέβαια δίκιο ο κύριο Ντομινίτσι ότι οι χώρε που βρίσκονται σε φάση εξυγένσης δεν θα πρέπει να αξιολογούνται πλέον. Θα πρέπει να ανακαλείται η αξιολόγησή του, διότι έχουν διαφορετικέ προοπτικέ. Αν δούμε τι διάφορες χώρες μάλιστα διαφέρουν μεταξύ του. Η Ιρλανδία τα πάει σχετικά καλά στα πλαίσια του προγράμματο εξυγένσης. Ε, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Ή εκεί οι επενδυτέ, τα άτομα, έχουν δικαίωμα να αντλούν τα δικά του συμπεράσματα για την πορεία των διαφορών χωρών και το πώ προχωρά το πρόγραμμα ανάκαμψη τη οικονομία του. Επίση, οι επενδυτέ βρίσκουν τις αξιολογήσεις χρήσιμες ε, για να λάβουν αποφάσει, καταλαβαίνοντα ποια είναι τα πιο επικίνδυνα χρέη, διότι οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν τις ε, κινήσεις της αγοράς. Εάν ε, περιθμίσουμε το χώρο αυτό, ουσιαστικά θα αποφύγουμε να υπάρξουν νέοι συμμετέχοντε στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ καλά τι προτάσει θα γίνουν και να καθορίσουμε από κοινού του στόχου που θέλουμε να πετύχουμε. Ανυπομονώ για τη συνεργασία με του συναδέλφου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πασκάλ. Ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο για ζητήματα που ούτως ή άλλως σχολιάστηκαν προηγουμένω από τους συναδέλφου. Αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε στην ε, ουσία του θέματος. Κατευθείαν, και αυτό είναι πολύ καλό. Για τη σύγκρουση των συμφερόντων, κατά πρώτο. Συμφωνώ με τον Ζαν ε, Πολ ότι θα πρέπει να περάσουμε από το πρότυπο του πληρωμή από τον εκδότη ε, στην πληρωμή από τον επενδυτή. Σήμερα Υπάρχει σαφώ σύγκρουση συμφερόντων, όπω το πρώτο που έχει διαμορφωθεί. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να καθορίσουμε ένα ενδιάμεσο σύστημα. Ένα σύστημα που να μοιάζει με διαγωνισμό. Να υπάρχει δηλαδή ένας μεσάζων μεταξύ του εκδότη προϊόντος, αυτού που προσφέρει το προϊόν, το προϊόν και του επενδυτή αλλά ούτε ο εκδίδων, ούτε ο επενδυτή, να πληρώνουν ουσιαστικά τον λογαριασμό απευθεία, για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αφύνδρομη. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια προμήθεια. Προμήθεια η οποία να λαμβάνεται και από τον επενδυτή και από τον εκδίδοντα και η οποία τελικά να καλύπτει τους οργανισμούς που αξιολογούν τα προϊόντα αλλά να μην υπάρχει εμπορικός συσχετισμό μεταξύ του οίκου και του επενδυτή του οίκου και του εκδίδοντα του προϊόν. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν να λειτουργεί με βάση ένα διαγωνισμό μεταξύ όλων των οίκων που λειτουργούν ε, στην αγορά και όχι μόνο των μεγαλύτερων. Αυτό θα μπορούσε να έχει και δημόσιο χαρακτήρα, κρατικό δηλαδή, βάσει του προτύπου που είχε προτείνει και το Κοινοβούλιο στην εποχή της έκθεσης Κλίντς. Δηλαδή όχι κάτι που να το κατευθύνουν τα κράτη, προφανώς. Γι' αυτό και δεν είμαστε υπέρ του να υπάρχει ένας κρατικός ε, οίκος ε, δημόσιου χαρακτήρα φορέας. Καλύτερα να υπάρχει κάποιο ίδρυμα, ίδρυμα με διακυβέρνηση ανεξάρτητη, άσχετη από τα ιδιωτικά συμφέροντα υπό την αυστηρή έννοια, αλλά και από τις κυβερνήσεις το ίδιο. Αυτός προς την πρόταση που θέλαμε να σας κάνουμε και να την εξετάσουμε όλοι μαζί για να βγούμε από το σημερινό μοντέλο, το πρότυπο και να αποφύγουμε κάθε τέτοιου είδου προβλήματα ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων. Έπειτα για την ΕΣΜΑ. και την ε, λεγόμενη, τον λεγόμενο εναρμονισμό των ε, προτύπων. Δεν συμφωνώ με το συμπέρασμα ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να κυρώσει το πρότυπο που θα επιλέξουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή το κυρώνει το εγκρίνει, ότι αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε ανερμόνιση. Απλώς ε, σημαίνει ότι είναι ένα μοντέλο που μπορεί να λειτουργεί. Ότι φταίει λογικά μπορεί να κάνει για εκείνη τι δικέ τη συστάσει, αλλά δεν σημαίνει ότι κύρωση μοντέλου ισοδυναμεί με τέλεια λειτουργία του μοντέλου. Υπάρχουν πολλά μακροοικονομικά μοντέλα που διαφέρουν μεταξύ του. Κάποια είναι φιλελεύθερα, κάποια άλλα όχι, τη μια ή τη άλλη οικονομική ε, φιλοσοφία. Μπορεί να είναι και τα μεν και τα δε αλλά δεν δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Ε, το να στοχεύουμε λοιπόν την εναρμόνιση δεν νομίζω ότι είναι ο στόχο, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει εξίσωση μεταξύ κύρωση του μοντέλου, έγκριση και ε, τη εναρμόνιση. Εδώ. Για το θέμα των ε, αξιολογήσεων και των συστάσεων που γίνονται. Ποιο είναι ο ρόλο των οίκων πιστοληπτική αξιολόγηση να αξιολογούν το βαθμό του κινδύνου. Όπω είπε και ο συντηρητικό συνδέλφο, αυτό που κάνουν είναι ότι αντικατοπτρίζουν τα αισθήσει που υπάρχουν στην αγορά. Το market sentiment, όπω θα λεγόταν. Ε, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό κάνουν μόνο. Το είπατε, έτσι. Το είπατε. Αυτό ακριβώ μπορούμε να του καταλογίσουμε. Ότι η αξιολόγησή τους δεν είναι αναγκαστικά εύστοχη. Ουσιαστικά απεικονίζουν το τι κάποια δεδομένη χρονική στιγμή ε, αισθάνεται η αγορά, φαίνεται να συμβαίνει στην αγορά. Όπως η Ιρλανδία που κάποια στιγμή μπορεί να φαίνεται αξιόπιστη και τελικά μετά από λίγο μπορεί να δείχνει ότι θα πτωχεύσει ή για την Ελλάδα το αντίστροφο. Δείχνουν λοιπόν το τι τάσεις επικρατούν στην αγορά κάποια δεδομένη στιγμή. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τον, κυκλικό χαρακτήρα των οικονομικών φαινομένων. Και επιτρέπουν στους επενδυτές να δουν αν θέλουν να διακινδυνεύσουν ή όχι. Όμως νομίζω ότι η συνολική λειτουργία στο οικονομικό σύστημα είναι να αξιολογούν κινδύνους. Δεν βλέπω γιατί αυτή η λειτουργία θα πρέπει να τους οδηγεί να κάνουν και συστάσεις. Να δώσω δύο παραδείγματα. Σήμερα η οίκη επιστολητικής αξιολόγησης έχουν ακριβώς το εξή αίτημα από την Ευρωζώνη να γίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοραστή των κρατικών ομολόγων. Και ο, τελευταί, ο ουσιαστικός δανειστής, εφόσον χρειαστεί, αν διαβάσετε όλα τα έγγραφα της Standard Poor's και της ε, Fitch, θα το δείτε, της Moody's μάλλον, θα το δείτε αυτό. Ε, Όμω άλλο είναι να γίνονται συστάσει. Μπορεί να πει ένα οίκο προστολεπτική αξιολόγηση ότι υπάρχει πρόβλημα, να το εντοπίσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει συστάσει. Μπορεί να πει για τι συντάξει, για το συνταξιοδοτικό, ότι υπάρχει δέσμευση των τόσων δι ευρώ από την πλευρά του κράτου που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται. Αυτό είναι αξιολόγηση κινδύνου. Τώρα, το κατά πόσο είναι ε, θεμητό ο αναλυτή τη Standard Poor's ή τη να λέει ότι στα 67 πρέπει να πάει το συνταξιδοτικό όριο, περισσότερε εισφορέ, ε, περισσότερα έσοδα για τι συντάξει ή ΦΠΑ για τι επιχειρήσει για να πάνε στι συντάξει, αυτό είναι ζήτημα πολιτικών αποφάσεων, δημοκρατία. Δεν μπορεί να τι ε, συστήνουν οι πιστολεπτικέ αξιολογήσει. Αυτά λοιπόν να τα σκεφτούμε τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κινδύνου, τι αφορά την μεθοδολογία και τι έχει να κάνει με την ε, πολιτική ιδεολογία. Αυτό δεν έχει καμία ε, σχέση εδώ με το θέμα μας. Δεν λέω ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο ένα ιδεολογικό μοντέλο που να επικρατεί, ούτε ότι αυτό που αντίκειται στις δικαιοθάτικα μου τα πιστεύω είναι λανθασμένο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το ζήτημα κατά πόσο νομιμοποιούνται οι επιστολοπτικές αξιολόγησεις να κάνουν πολιτικές συστάσεις. Και μια πρώτη τελευταία παρατήρηση. Η εξάρτηση και οι ρυθμίσει σε σχέση με τη λειτουργία των εικόνων. Θα πρέπει να αποφύγουμε οι επενδυτέ να αναγκάζονται να πουλήσουν του τίτλου όταν αλλάζει ο βαθμό και περνάει από το τριπλό Α στο διπλό, ή τέλο πάντων ότι υπάρχει μια υποβάθμιση. Θα πρέπει να φροντίσουμε με το κείμενο να μην υπάρχει τέτοια επιρροή. Δηλαδή, αν κανεί έχει αγοράσει Μάλλον, να διαχωρίσουμε τα πράγματα ω εξή. Να λέμε, είναι κανεί υποχρεωμένο. Μάλλον, εάν ο κανόνα ε, επιβάλλει την αγορά τίτλων 3α για την απόλυτη ασφάλεια, αυτό να ισχύει, αλλά το εάν το προϊόν που αγοράστηκε με τριπλό α υποβαθμιστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανεί υποχρεωμένο να το πουλήσει. Γιατί έχει τουλάχιστον μια διάρκεια, μια κάλυψη για ένα χι αριθμό ατών. Μην ε, σκεφτόμαστε δηλαδή με βάση την ε, fair value, όπως, γιατί αυτά είναι συζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύκλο των οικονομικών φαινομένων, όπως γίνεται με την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει βεβαίω να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ μας για να προχωρήσουμε σε αυτό. Και τέλος, σε σχέση με το Ίδρυμα. Το έχω ήδη σχολιάσει και συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό που προτείνει η έκθεση Κλίντ. Θα πρέπει βεβαίω να αναζητήσουμε και την πλειοψηφία εδώ, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει ούτε ιδέε για το ίδρυμα, ποια θα είναι η σύνθεσή τη, η διακυβέρνησή τη. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτήν την ιδέα και να σκεφτούμε, να βρούμε ένα μοντέλο που να μην είναι ούτε το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ίδρυμα ή να δούμε τι θα μπορούσε η αγορά ίδια να ζητήσει ως δημόσιο φορέα που να εξυπηρετεί και το οικονομικό σύστημα. Πάντως, ιδίως για τις επιχειρήσεις, το να υποχρεώνουμε τι οίκου πιστοληπτική αξιολόγηση να λαμβάνουν του έξω οικονομικού παράγοντε υπόψη για τον κίνδυνο, ιδίω του περιβαλλοντικού, αυτό σήμερα μα φαίνεται απαραίτητο. Το είδαμε με την BP λόγου χάρη ε, είναι ένας κίνδυνος που κανείς δεν, λαμβάνουν ε, υπόψη, που κανείς δεν λαμβάνει υπόψη. Σημαντικό είναι λοιπόν να συνυπολογίζεται για να υπάρχει μια περισσότερο σφαιρική εικόνα του κινδύνου για τους ε, μετόχους, τους επενδυτές, διότι οι περιβαλλοντικές απειλές μπορεί να έχουν σοβαρέ οικονομικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε με τους κοιόδης εισηγητές. Έχουμε περίπου μισή ώρα μπροστά μας. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε αυτή τη συζήτηση. Έχω ακόμη τέσσερι ομιλητέ. Ρενάλντο, μάλλον θα θέλει απαντήσει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπω συντομότεροι από ότι. Να είστε κάπω συντομότεροι από ό,τι όλοι. Υπάρχουν κι άλλοι. Όλοι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο για την Επιτροπή. Τους δόθηκε ευκαιρία να δουν την έκθεση. Θα δούμε πώ θα πάει. Εάν μπορούν να είναι σύντομοι συνάδελφοι στι παρατηρήσει του, ίσω να μείνει χρόνο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόμα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ο Ζαν είχε ζητήσει να τον αξιολογούμε συνέχεια. Σου δίνω τριπλό αλφα, Ζωάν Πολ. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται με τους οίκους αξιολόγησης. Έχει υποβαθμιστεί η Ιταλία και η Ισπανία, ακόμα και το Βέλγιο πρόσφατα. Οι φορείς λοιπόν αυτή η αξιολόγηση. Γιατί είναι τόσο λανθασμένη η ιδέα του να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης αν είχαμε ένα φορέα ο οποίος ήταν πραγματικά ανεξάρτητος που να χρηματοδοτείται από τα κράτη αλλά είναι ανεξάρτητος και δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούμε να το έχουμε. Λέμε ότι οι τρεις οίκοι ελέγχουν τα 95% της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό οδηγεί σε πολλά προβλήματα στις ε, διασυνδέσεις τους και την εξάρτηση από αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι σωστό το να λέμε όμως ότι όλα αυτά τα οποία γίνεται είναι απλώς η άποψη των εταιριών αξιολόγησης. Είναι και μια πολιτική κρίση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι έχουν συνολικό τζίρο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στι ΗΠΑ Πολιτείες πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να πούμε ότι θα πρέπει εφόσον παίρνουν τόσα πολλά λεφτά να έχουν και ευθύνη για τις κρίσεις τις οποίες εκφέρουν. Υπάρχουν, όπως είπε και ο Βολφ Κλίντς, μικροί περιφερειακοί και εθνικοί φορείς σε εθνικό επίπεδο. Γιατί να υπάρχουν αφού δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να λαμβάνεται υπόψη η θέση τους και η άποψή τους. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις ε, μετοχές των φορέων ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Warren Buffett έχει 25% των μετοχών σε αυτές τις εταιρείες. Επομένως δεν μπορεί να είναι αδιάφορο σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκού χρέους. Έχει δίκιο ο Wolf Θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία η οποία απαιτεί την αξιολόγηση από αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους φορείς αξιολόγησης. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταγράψουμε αυτό σε και να το διατηρήσουμε στην αιώνιότητα. Οι νόμοι και οι νομοθετικέ διατάξει έχουν ένα χρόνο ζωή. Δεν πρέπει να εξαρτώμεθα μόνιμα από αυτέ τις, αυτές τις ε, εταιρείε αξιολόγηση. Δεν πρέπει να τι απαγορεύσουμε, αλλά πρέπει να υπόκεινται σε μια ρύθμιση. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά θέματα όπου λέμε ότι αυτά δεν είναι σημαντικά για τους απλούς ανθρώπους. Όχι, εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό θέμα το οποίο είναι θέμα εξουσίας και έλλειψης εξουσίας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης και την προηγούμενη φορά είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Τα βασικά προβλήματα όμως δεν έχουν τροποποιηθεί. Είναι περισσότερο από ποτέ κατεπήγον να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα συμφωνούσα γενικά με αυτά που είπατε, ότι ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρξει κάποιος βαθμός ανταγωνισμού, ώστε κανένας συγκεκριμένος παίκτη να μην ελέγχει όλη την αγορά. Αυτή είναι και η ηθική βάση της οικονομίας της αγοράς, ότι κανένας από τους συμμετέχοντες στην αγορά δεν έχει απόλυτη εξουσία. Εδώ πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων, ίσως εκτός της άκρας αριστεράς. Αλλά θα έπρεπε όλοι να συμφωνούμε γι' αυτό και με εντυπωσιάζουν κάποια σχόλια που κάνανε ορισμένοι. Αν συμφωνούμε για αυτό το στόχο, τότε δεν θα έπρεπε να υποστηρίξουμε κάποια λύση σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι εδώ έχουμε ε, παίκτες στην αγορά που έχουν κυριαρχική εξουσία. Καμία λύση λοιπόν που θα υποστηρίξουμε δεν θα πρέπει να τους αφήνει να διατηρούν αυτή την υπερβολική εξουσία. Εφόσον υπάρχει υπερσυγκέντρωση, όπως είπε Στόμας, όταν υπάρχει υπερσυγκέντρωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ανταγωνισμού και να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτά τα καρτέλια, αυτές τις συνενώσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους, γιατί η διάσπαση είναι κάτι το οποίο είναι μια ομή και απότομη διαδικασία και δεν είναι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή ως νομοθετών. Είναι άλλοι οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο και κανονικά είναι στο χέρι της Κομισιόν να το πράξουμε. Αυτό όμως το οποίο εμεί θέλουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μια αριθμιστική εξουσία για να μειώσουμε και την δύναμή τους στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα ευρωπαϊκού χαρακτήρα για αξιολόγηση. Συμφωνώ με αυτού που είπαν ότι δεν πρέπει να είναι ένα δημόσιο σώμα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον, αλλά δεν πρέπει να είναι δημόσιο φορέα. Α επανέλθουμε λοιπόν <clears throat> στην αρχική μα πρόταση και να την εγγράψουμε στην νομοθεσία. Δεύτερον, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όσο εξακολουθούν να υπάρχουν δεσπόζουσε εταιρείε στην αγορά αξιολόγηση, θα πρέπει τουλάχιστον να περιορίσουμε την εξουσία του. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μεγάλο χρηματοπιστωτικό φορέα που μπορεί να κάνει τη δική του αξιολόγηση κινδύνων, δεν θα πρέπει να τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις απόψεις των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Γιατί τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης των τραπεζών και των πιστοτικών ιδρυμάτων βασίζονται στους οίκους αξιολόγησης. Αν επενδύει τα χρήματά του σε μια τράπεζα ή αγοράζει κάτι στο ίντερνετ, το αγοράζει μόνο επειδή κάποιο έθεσε ένα τριπλό α στην αξιολόγηση αυτού του προϊόντος. Όχι, πρέπει ο καθένας να κρίνει από μόνος του. Οποιοδήποτε φορέας της αγοράς που έχει ένα τουλάχιστον κρίσιμο μέγεθος θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δική του αξιολόγηση. Επομένως, θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από την υπερβολική εξάρτηση από τους φορείς αυτούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Συμφωνώ με αυτό που λες ότι ένας μικρός χρηματοπιστωτικό παίκτη μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει μόνο σε ένα πολύπλοκο προϊόν. Αλλά πάνω από ένα κατόφλι μεγέθου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόνομη αξιολόγηση και θα πρέπει να επιτρέπεται να κάνει αναφορέ <clears throat> στου φορεί πιστοληπτική αξιολόγηση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση που το κάνουμε αυτό, τους δίνουμε με την ομοθεσία μας ήδη ακριβώς την εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν σε μια οικονομία της αγοράς. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε αυστηρότερους κανόνες πέραν αυτού ένιωσα έκπληξη γιατί πολλοί είπαν ότι δεν πρέπει να έχουμε μία εναλλαγή επιβεβλημένη των τριών φορέων αξιολόγηση, αλλά δεν πρότειναν κανένα μέτρο για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα να παροτρύνω όλε τι πολιτικέ ομάδε να αναπτύξουν προτάσει για το πώ μπορούμε να σπάσουμε την υπερβολική εξουσία αυτών των φορέων. Δεν μπορεί να λέει κανεί είμαστε εναντίον τη εξουσία του, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική εναλλαγή. Βρείτε λοιπόν, σας παρακαλώ, κάποιο τρόπο να σπάσουμε αυτή την υπερβολική εξουσία που δεν έχει ρόλο να παίξει στην οικονομία της αγοράς. Και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η κατάσταση. Έχουμε κράτη τα οποία έχουν αναλάβει τα ρίσκα που πήρανε οι ιδιωτικές τράπεζες για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Δίνουμε τη δυνατότητα στις ιδιωτικές αυτές εταιρείες αξιολόγηση να έχουν ένα μονοπόλιο υπονομεύουμε, υποσκάπτουμε την ηθική βάση και τη δημόσια υποστήριξη για μια οικονομία αγοράς. Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την κατάχρηση της οικονομίας της αγοράς που δεν έχει καμία σχέση με μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Σας παρακαλώ, ακούστε αυτά τα οποία ζητούν οι πολίτες που θέλουν να σπάσει αυτή η εξουσία των αξιολόγησης και που είναι μια αίτηση που συνάδει με ένα κράτος δικαίου και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Δεν αρκεί λοιπόν να πούμε όχι σε αυτό το μέτρο ή σε κάποιο άλλο μέτρο. Θα πρέπει να δράσουμε και θα πρέπει να βρούμε πιστικές λύσεις. Συγγνώμη συνάδελφοι, δεν μπορούμε ομιλητά. Ο Πίτερ Ζήμων έχει το λόγο τώρα. <coughs> Για ένα σημείο θα ήθελα να σταθώ το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και ο, Βόλφ ο, αναφέρθηκε. Το θέμα της δομής ε, ιδιοκτησίας των ε, φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης και των ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων. Από αυτό που βλέπω στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Έχουμε αυστηρές ε, προδιαγραφές σε νομικό επίπεδο για τα πιο μικρά ε, θέματα για τις πιο μικρές ε, επαγγελματικές ομάδες για να αποφύγουμε τις συγκρίσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων για τους δημοσιογράφους, για τους επικεφαλής διοικητικών συμβουλίων, για όλους αυτούς οι οποίοι φεύγουν από μία ε, εργασία και περνάνε σε ένα διοικητικό συμφέρον. Συμβούλιο. Μιλάμε για τους επιτρόπους, μιλάμε για τους πολιτικούς όταν φεύγουν από το αξίωμά τους. Για όλους αυτούς έχουμε μια μεγάλη ευαισθησία. Δεν έρχεται όμως για τους φορείς αξιολόγησης. Δεν έχουμε δείξει ενδιαφέρον για αυτό το πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων παρά το γεγονός ότι μας έχουν απασχολήσει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις συζητήσεις μας όλα αυτά. Και θα ήταν χρήσιμο η Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Τι λέει όμως η Κομισιόν αντί για κάτι τέτοιο. Καμία επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει μετόχους οι οποίοι ξεπερνούν το 10% ή έχουν μια σημαντική θέση σε αυτήν την ε, επιχείρηση η οποία ασκεί την αξιολόγηση. Αυτό αποκλείει τη συγκρούση συμφερόντων. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι. Τη σύγκρουση συμφερόντων δεν προκύπτει μονάχα από το γεγονός ότι ένας ε, ε, μέτοχος σε μία εταιρεία αξιολόγηση είναι συγχρόνω και μέτοχος στην αξιολογούμενη εταιρεία. Αυτό δεν φτάνει <clears throat> για να αποκλείσει ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό συμφέρον σε σχέση με το πόρισμα της αξιολόγησης. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει κερδοσκοπήσει σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της αξιολογούμενης εταιρεία. Αν από την πλευρά λοιπόν των μετόχων υπάρχει ένα συμφέρον να υπάρξει μια αξιολόγηση που πηγαίνει προς την α ή στη β κατεύθυνση και έχουμε μια δομή η οποία επιτρέπει όλοι οι μέτοχοι αυτοί να μπορούν να έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα γιατί όλοι παίζουν μέσα σε αυτό το χώρο τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και σας υπενθυμίζω αυτό που έκανε η Roland Becker, μια γερμανική εταιρεία, σε σχέση με τη μορφή των ε, συμμετοχών σε αυτές τις εταιρείες. Δεν είναι κάποιος που μπορούμε να τον υποψιαζόμαστε για ακραίο σοσιαλισμό. Δείχνει εδώ πέρα αυτή η αξιολόγηση ότι όλοι αυτοί έχουν ε, καταφέρει να βγάλουν λεφτά από τις αξιολογήσεις των εταιριών αξιολόγησης η BlackRock, η Goldman Sachs, όλοι αυτοί συμμετέχουν στο παιχνίδι με τις εταιρείε αξιολόγησης. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τις ε, συγκρούσεις συμφερόντων και να προσπαθήσουμε να τις αποτρέψουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο όπως έχουμε κάνει με όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων και ημών των ιδιών των πολιτικών. Καλώς έβαλα και τον εαυτό μου στον κατάλογο αγοριτών και για πρώτη φορά δεν θα βγάλω το όνομά μου προς όφελος των άλλων μελών και θα πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το πρόβλημα αυτό που έχουμε εξετάζοντας τη μεθοδολογία και πώς οι οίκοι αξιολόγηση λειτουργούν. Γιατί το λέω αυτό, διότι αναπόφευκτα διεξάγονται συζητήσει όταν ε, δημιουργείται κάτι ή όταν ελέγχεται ε, μια αξιολόγηση λέμε ότι το EFSF που θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι υποπτό ε, συζητάμε οίκους αξιολόγησης ε, σχετικά με τη δική του αξιολόγηση του EFSF και αυτό συνεχίζεται και από τη στιγμή που οίκος αξιολόγησης βάλει μια χώρα ή μια εταιρεία υποπαρακολούθηση ε, υποβάλλεται το ερώτημα προς τον οίκο αξιολόγηση γιατί το κάνατε αυτό και επιστρέφει η απάντηση λέγοντας ότι θεωρήσαμε ότι υπάρχει το τάδι δίνα θέμα. Δεν είμαι σίγουρη λοιπόν ότι είναι απαραίτητο σωστό να λέμε ότι αυτό αποτελεί πολιτική παρεμβολή όταν τους ρωτάμε γιατί κάνατε κάτι και είναι δημόσια μεθοδολογία. Είναι σωστό να λένε ανησυχούμε για την, το σύστημα το συνταξιοδοτικό σας ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά το ερώτημα έρχεται πώς θα αλλάζουμε αυτό. Είναι προφανές ότι αν κάνεις τις αλλαγές που ανησυχούν τους οίκους αξιολόγηση αλλάζει η αξιολόγηση. Έτσι λειτουργούν αξιολογηση αλλαζει ετσι λειτουργουν αυτα και πάντα τα στοιχεία θα είναι ιστορικά. Διότι πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες από τις αγορές και από διάφορα γεγονότα. Και όσοι συμμετείχαν μαζί μου σε άλλους τριμερείς διαλόγους θα γνωρίζει ότι πάντα επιμένω να έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερα στοιχεία πραγματικού χρόνου από διαφορετικές πηγές. πηγές συγγνώμη. γιατί, για να προχωράμε πιο γρήγορα. Και αν επιμένουν οι συνάδελφοι να αντιστέκονται σε αυτά που ζητώ, και αυτά που ζητάει η ΕΚΤ, τότε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Δεν θα έχουμε καλύτερη ανάλυση πραγματικού χρόνου χωρίς να βασιζόμαστε σε φορείς που θα πρέπει να συλλέγουν οι ίδιοι τα στοιχεία. Το να απαλλαγούμε από τι αξιολογήσεις είναι δύσκολο, το προσπαθούν στη ΣΥΠΑ και όταν ήμουν εκεί το συζήτησα. Και αισθανόταν οι Αμερικανοί ότι ε, εξέταζαν ε, το θέμα των swaps και λοιπά και δεν, δεν έβγαζαν άκρη. Το να εξαιρείται μια χώρα, υπάρχει αναστολή για μια χώρα που ακολουθεί πρόγραμμα διάσωσης, ίσως προχωράει πιο πολύ μακριά. Το έχουμε ξανακάνει αυτό όταν συζητήσαμε για τα ασφαλισμένα προϊόντα και λέγαμε αν θα έπρεπε να υπάρχει ένας στερίσκος και κάποια αναφορά στην αξιολόγηση που θα ξεχώριζε ένα περίπλοκο προϊόν από ένα πλούστερο. Και το να βάλουμε ένα σταρίσκο και να λέμε ότι η χώρα αυτή είναι σε εντό προγράμματο, ίσω είναι λογικό, αλλά αυτό που είπε ο Άσλεϊ Φόξ ίσω είναι σωστό. Θέλουμε να δούμε, υπάρχει κάποια πρόοδος που σημειώνεται και αυτό βοηθά. Κατηγοριοποίηση όμως που θα δείχνει ότι κάτι συμβαίνει που δεν είναι απόλυτα ομαλό, δεν ξέρω, ίσως να είναι εφικτό. Οι επενδυτές τα ρυθμίζουν αυτά και θέλουν και την αξιολόγηση από τους μεγάλους οίκους αξιολόγηση οι επενδυτές. Και ίσως πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Όπως και με τον έλεγχο, παρόμοιο το πρόβλημα. Μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν και υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να διορίσουν ελεγκτέ και πρέπει να κάνουν αξιολόγηση και αυτοί αισθάνονται ότι αν επιλέξουν μικρότερε εταιρείε ε, μπορεί να κατηγορηθούν αν πάνε στραβά τα πράγματα. Είναι σαν ταινία κάτσε 22. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Θα μπορούσα να πω περισσότερα, σταματήσω. Η Λίσσα είναι η επόμενη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Sharon. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μια κάποια αντίφαση μεταξύ της περιγραφής που κάνουμε για αυτό το οποίο είναι προφανές στην λειτουργία των οίκων ενώ συγχρόνως δεν αντλούμε όλα τα συμπεράσματα από τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό το οποίο λέει. Αν έχουμε μια αγορά η οποία κυριαρχείται κατά 95% από τρεις εταιρείες, Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διείσδυση συμφερόντων που αφορά την ε, αξιολόγηση και έχει να κάνει και με το κέρδος αυτών των εταιριών. Δεν έχουμε λοιπόν πληροφορίες που είναι ουδέτερες και προς το συμφέρον το δημόσιο. Έχουμε να κάνουμε με μια επιχείρηση που έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη δική της κερδοφορία. Αυτό είναι το εγχείρημα των εταιριών αξιολόγησης. Όλα αυτά σημαίνει ότι εμείς κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες στον τομέα του ανταγωνισμού και παραγνωρίζουμε μια σοβαρή κατάσταση στην οποία τρεις εταιρείε ελέγχουν όλη την αγορά. Όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν περιγράφουν το πρόβλημα και μετά υποχωρούν στις δικές τους μικρές προτάσεις για μια λύση. Τι θα κάνουμε για τη στρέβλωση ανταγωνισμού μόνο με το να εξασφαλίσουμε ότι αν κάποιος έχει υπερβολικό μερίδιο της αγοράς θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν το οπλοστάσιο που έχουμε σε, στα πλαίσια του ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείε. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να γίνονται πράγματα τα οποία τα απαγορεύουμε στην πολιτική ανταγωνισμού έχουμε πει ότι πρέπει να μειώσουμε τα υπερβολικά μερίδια της αγοράς, να μειώσουμε και να καταλύσουμε και τα φράγματα εισόδου στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Βολφ Κλίνς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει και κάποια διαφάνεια για την ε, μετοχική δομή των εταιριών αυτών. Πρέπει λοιπόν η πολιτική ανταγωνισμού να μπει στο παιχνίδι αυτό με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα σοφέ και να αρθρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπεραστεί αυτή η υπερβολική εξουσία που κάνει μια ολόκληρη αγορά να είναι το ιδιωτικό γήπεδο τριών εταιριών αξιολόγηση. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί επαρκώ η πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί και συμφωνώ με τα περισσότερα τα οποία ελέγχθηκαν, ιδίω για το γεγονό ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ουσιαστικά έχει αναγνωρίσει σε ρυθμιστικό επίπεδο αυτές τις ίδιες αξιολογήσεις των οίκων που αυτή τη στιγμή εμείς επικρίνουμε. Τέλο, θέλω να πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό ότι ορισμένε χώρε κάτω από ορισμένε συνθήκε δεν μπορούν να προχωρήσουν στις προσπάθειές τους γιατί οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγηση είναι προφητείες οι οποίες αυτοεκπληρούνται ουσιαστικά και με τον τρόπο αυτό μπορούν να κάνουν την αγορά να λειτουργεί έτσι ώστε να επαληθευτούν οι δικέ του προβλέψει. Αυτό σημαίνει υπερβολική εξουσία των εταιριών αξιολόγηση. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Δεν χρειάστηκε τα 7 λεπτά η Λίζα. Ήταν αυτή και εκείνη που κάναμε. Συμπληρώσαμε τα 7. Όλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιούμε περισσότερο στα CDS από τις ε, αξιολογήσεις αυτή θα είναι μια νέα έκθεση του Πασκάλ. Για να περιοριστεί η εξουσία της αγοράς. Ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι οι χώρες και η πολιτική των χωρών, συμπεριλαμβανόμενοι ημών, να συμπεριφερόμαστε σωστά. Έτσι περιοριζόμαστε την εξουσία της αγοράς. Αν δεν πιστεύετε στους οίκους αξιολόγησης, θα πιστεύετε το διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά που είπε στις Financial Times εχθές, είπε ότι όλοι οι οίκοι έχουν δίκιο όσον αφορά τα κρατικά χρέη. Και αυτό είναι το δυσκολότερο. Να πυροβολείτε τους υπεύθυνους, όχι μόνο τους πιανίστες. Τώρα σοβαρά. Είναι μια πρόταση που θα πρέπει να επεξεργαστούμε και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που αν εισαχθούν θα κάνουν πιο ευάλωτη την αγορά. Δεν συμφωνώ με τον Wolf Klims. Νομίζω ότι κάποιες προτάσεις δεν θα είναι επωφελείς για την επίτευξη των στόχων μας. Προσπαθήστε να είστε κάπως προσεκτικοί. Μη λησμονείτε ότι παρόλο που οι οίκοι αξιολόγηση δεν τα πήγαν καλά στη ΣΥΠΑ, έκαναν λάθος, οι πολιτικοί τους έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά τα σφάλματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Διέγκο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή δουλειά στον εισηγητή μας για αυτό το θέμα που δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, έχουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για το εγχείρημα αυτό, γιατί είναι η τρίτη μεταρρύθμιση αυτού του νομοθετήματος, κάτι το οποίο δημιουργεί και αβεβαιότητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, ευκαιρία για να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό και όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένο σε σχέση με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτή την πρόταση του εισηγητή. Υπάρχουν σημεία για τα οποία έχω κάποιες αμφιβολίες και κάποιες παραλήψεις. Για τα θετικά ε, στοιχεία είναι αυτό που λέει ότι πρέπει να εξαλείψουμε τις νομοθετικές αναφορές στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης για να ξεπεράσουμε την υπερβολική εξάρτηση και να μπορούν και να πρέπει οι επενδυτές να κάνουν από μόνοι τους την αξιολόγηση κινδύνου. Γιατί ό,τι κάνουν οι εταιρείε αξιολόγηση μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι οι επενδυτές. Επίσης, να υπάρχει αυτονομία στην αξιολόγηση και τέλος το θέμα των ειδικών κανόνων σε σχέση με το κρατικό χρέος, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα αυτό. Τώρα, τα σημεία στα οποία έχω αμφιβολία μετά από μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου του εισηγητέ. Καταρχήν το θέμα να μην μπορεί να υπάρχει συγχώνευση μέσα στα 10 χρόνια των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης παρά το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα, θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών συγχωνεύσεων και εξαγορών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, η δημιουργία του μοντέλου υποχρεωτικής αναλλαγής που αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους. Φοβάμαι ότι μια τέτοια αναλλαγή θα εξυπηρετήσει μονάχα να υπάρξει καλύτερη κατανομή της αγοράς μεταξύ των τριών αυτών φορέων αξιολόγηση. Δεν πρόκειται να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν θα δημιουργήσει τις καταστάσεις για να μειωθεί η εξουσία αυτών των φορέων, μάλλον θα μειωθεί ο ανταγωνισμός. Επίσης, η Κομισιόν έχει προτείνει μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 να προτείνει ένα νέο μοντέλο για την, ε, για την αξιολόγηση, για την αμοιβή των εταιρείων αξιολόγησης, όχι μονάχα δηλαδή από τον εκδότη, αλλά και από άλλους φορείς. Μας ενδιαφέρει εδώ να εξασφαλίσουμε μία σταθερότητα σε νομικό επίπεδο για, την, ε, ε για τα θέματα αυτά και επίσης η έκθεση, η θέση της Κομισιόν δεν δέχεται τη δυνατότητα να υπάρξει μια δημιουργία Ευρωπαϊκού Φορέα Αξιολόγησης με δημόσια χρηματοδότηση αλλά ε, ανεξάρτητη. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εταιριών αξιολόγησης που λειτουργούν παρόλα αυτά ήδη σήμερα. Αυτό θα ήταν μια καλή λύση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού. Η Κομισιόν επίσης θεωρεί ότι το κρατικό χρέος θα πρέπει να είναι εκτός του συστήματος αυτού. Εγώ θέλω να επιστήσω εδώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι η, αξιολόγηση που γίνεται για κράτη τα οποία βρίσκονται σε προγράμματα εξυγίανσης δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί έτσι κι αλλιώς οι χώρες αυτές δεν συμμετέχουν στις αγορές για τη χρηματοδότησή τους, επομένως αυτές οι αξιολογήσεις δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε τώρα στον εισηγητή. Φοβούμαι δεν έχουμε χρόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουν πολλά να πούν τα μέλη και δεν μπόρεσα να δώσω το λόγο. Θα προτιμούσα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντί για σας να κλείσουν εκείνη τη συζήτηση. Ωραία. Ο εισηγητή μας λέει καλύτερα να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πολύ τυχεροί. Ευχαριστούμε για την κυρια ντομενητη Ντομένιθη. Μια-δυο παρατηρήσεις προς απάντηση των σχολείων που έγιναν πολύ αναφέρθηκαν στο issuance payment model αντί για το να πληρώνει ο επενδυτής. Εδώ υπάρχει έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Αναφέρθηκε και αυτό το πρωί, νωρίτερα. Να δούμε το issuer pays model με προσοχή και το τι συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν εξαιτία από του μοντέλου και δεδομένων των εξελίξεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ γιατί και εκεί το εξετάζουν το θέμα αυτό. Για τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται. Εδώ ίσως υπάρχει μια παρανόηση για το τι ακριβώς προτείνει η Επιτροπή. Εάν με επιτρέπετε, πολύ σύντομα να εξηγήσω. Αυτό που προτείνουμε είναι η διάταξη σχετικά στον κανονισμό CRA, στο άρθρο 8 3, όπου λέγεται ότι ο οίκο αξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογία που να είναι αυστηρή, συστηματική, διαρκή, υποκείμενη σε κύρωση και σε ιστορικά στοιχεία δεδομένων των ε, αναδρομικών ε, δοκιμών, αυτό τι σημαίνει ότι η ΕΣΜΑ πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από τους οίκους συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσει. Δεν δίνουμε επιπλέον εξουσίε στην ΕΣΜΑ ώστε να κυρώνει επισήμω τι μεθοδολογίε ή να τι εναρμονίζει. Όχι. Του δίνουμε την. Τους φορτίζουμε με το καθήκον να ελέγχουν κατά πόσο συμμορφώνονται οι μεθοδολογίε με τι υπάρχουσε νομικέ υποχρεώσει. Όχι με νέε υποχρεώσει, με τι φυστάμενε. Το θέμα της υπερβολικής εξάρτησης αναφέρθηκε από, πολλές, από πολλούς παρεμένοντες είναι σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της όλης πρότασης. Έχουμε ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα πέρυσι το καλοκαίρι όταν προτείναμε το CRD4 όπου ζητήσαμε να περιοριστεί η εξάρτηση από τις αξιολογήσεις αυτές. Τώρα κάνουμε ένα δεύτερο βήμα με το πρόγραμμα αυτό ώστε να περιορίσουμε την εξάρτηση και με τους ΣΕΚΑΒ και με την οδηγία FMD και θα έχουμε και περαιτέρω προτάσεις για να περιοριστεί αυτή η, αξιολόγηση, η εξάρτηση από τις αξιολογήσεις και στον τομέα των κρατικών χρεών. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά ζητούμε από όλες τις αρχές ε, ελεγχού της ΙΖΑ και της ESRB να μην ε, κάνουν μία των ε, αξιολογήσεων στις κατευθυντήριες γραμμές τους. Θέλουμε να περιορίσουμε αυτή την αυτόματη εξάρτηση από τις αξιολογήσεις και στο επίπεδο της νομοθεσίας και το ευρωπαϊκό και κυρίως τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμοδίων αρχών. Τέλος, αναφέρθηκε ο κανόνας της εναλλαγής. Ε, καταλαβαίνω ότι πολλοί ε, βουλευτές έχουν ε, αμφιβολίες για το κατά πόσο αρμόζει και είναι εύστοχος ένας τέτοιος κανόνας. Από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας τέτοιος κανόνας τι θα σήμαινε κατά κύριο λόγο. Θα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις συμφερόντων προκαλεί το μοντέλο του issuer pays. Εδώ Θέλουμε λοιπόν να προλάβουμε τι συγκρούσει που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ε, πολιτών των προϊόντων και των ε, οίκων αξιολόγηση. Τώρα η αναλλαγή ανά τριετία ή σε μερικέ περιπτώσει ανά εξαετία ή περίοδο cooling off ε, για μια τετραετία. Αυτά ίσως να επέτρεπαν μια περισσότερη, περισσότερο δυναμική κίνηση της αγοράς, κάτι που είναι και μεταξύ των στόχων μας. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε κάποια μαγική λύση εδώ βέβαια για όλα τα προβλήματα. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις ιδέες του Κοινοβουλίου. είναι κάτι που μας ανησυχεί. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό της έλλειψης επιλογής και του περιορισμένου ανταγωνισμού στην σχετική αγορά. Και πάλι ευχαριστώ στον κύριο Ντομένιτση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λεωνάρντο, θες να πεις ένα-δυο λόγια. Απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να συζητήσουμε. Απλώς μία παρατήρηση. Το γεγονός ότι μπορεί μια απάντηση να θεωρείται εσφαλμένη ή να υπάρχουν διαφωνίες ως προς αυτήν, δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται κατά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους να παραδεχτούν ότι αντικειμενικά υπάρχουν προβλήματα και παρακαλώ να συμβάλλουν με τις εναλλακτικές τους ενδεχομένως προτάσεις ώστε να βρεθούν λύσεις. Um, Ευχαριστώ. πολύ. Θα γίνει μια κρόση στις 24 Ιανουαρίου. Το σχέδιο εκθέσεως θα πρέπει να είναι έτοιμο 28 Φεβρουαρίου, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 22 Μαρτίου. Προχωράμε τώρα σε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και θα επανέλθω σε λίγο με τον Υπουργό. Υπότιτλοι Okay, everybody. Λοιπόν, να πάψουν οι συζητήσεις και να καθίστε παρακαλώ. Και αν θέλετε να μείνετε, ας βγείτε ήσυχα παρακαλώ. Καθίστε. Ξεκολουθούν οι κουβεντούλες. Παρακαλώ εκτός ηθούσης. Αν θέλετε να ξαναέθετε στην Επιτροπή αυτή, δεν θα συζητάτε μέσα, εκτός. We have a time schedule. Right. Um... Right. We, we, as I'm sure... Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, φτάνουμε προς το τέλος της Πολωνικής Προεδρίας και ως ήθιστε θα διεξαχθεί άλλη μια ανταλλαγή απόψεων με τον Γιάζε Κροσόφσκι, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκοφήν. Θα του δώσω το λόγο περίπου για ένα δεκάλεπτο για να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την Προεδρία. Μετά θα ακολουθήσει και περίοδος υποβολής ερωτήσεων και απαντήσεις. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάρων. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να επικεντρωθώ επί των σημαντικότερων γεγονότων της Προεδρίας, όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον, και πώς συμβάλαμε εμείς στη διαμόρφωσή τους. Δεν τα ξεκινήσαμε πολύ άσχημα. Uh, Απευθύνοντας έκκληση τον Ιούλιο, ζητώντας σημαντικότατη μείωση των επιτοκίων, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των χωρών που είναι σε προγράμματα στους Ευρωζώνης, δηλαδή Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Κάτι που ελήφθη υπόψη γρήγορα, δεν το πέτυχε η ίδια η Προεδρία, ήταν απόφαση της Ευρωζώνης, αλλά ήταν δική μας πρωτοβουλία και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική, διότι τα προηγούμενα επιτόκια ήταν πολύ υψηλά ε, και έσπρωχναν τις χώρες προς παγίδα χρέους, τις προβληματικές χώρες Χαιρόμαστε λοιπόν που αυτή η πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή από τις χώρες Ευρωζώνης. Δεύτερον, επίτευγμά μας μαζί σας, βέβαια, βασιζόμενοι επί της άριστης δουλειάς της Ουγγρικής Προεδρίας, καταφέραμε συμβιβασμό επί του six που τείνουν να το υποτιμούν τώρα που υπάρχουν και άλλες ιδέες που ρίχνονται για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Γεγονός είναι ότι αν εφαρμοστεί σωστά η δέσμη των έξι μέτρων θα εξασφαλίσει ότι δεν θα επιστρέψουμε στην ε, φοβερή θέση που είμαστε σήμερα Α, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πλευράς οικονομικής. Ε, βέβαια, αφήνει αυτό, αυτό που γνωρίζαμε πολύ καλά ότι θα ήταν η βασική μας ανησυχία. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης του κρατικού χρέους και να βγούμε από αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφέρω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο. Βοήθησε πολύ όσον αφορά τον προπολογισμό του 2012, αν λάβει κανείς υπόψη τις παρούσες εντάσεις που υπάρχουν και, τις, και στις παγκόσμιες αγορές και στις αγορές κρατικού χρέους θα ήταν ε, πολύ επιβλαβές να είχαμε την ίδια ε, τα ίδια προβλήματα και αντιδικία που είχαμε το 2011 και ευχαριστώ πολύ το Κοινοβούλιο για την επικοδομητική στάση του. Κάτι πολύ σημαντικό που αντιμετωπίσαμε έλαβε χώρα τον Οκτώβριο το πακέτο επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ο Μάριο Ντράγκη, από ό,τι ξέρω, ήταν εδώ χθες και συμμερίζομαι αυτό που είπε, ότι παρόλο που το πακέτο ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών ήταν καλά σχεδιασμένο σαν σχέδιο, και περιέχει πολλές ε, διατάξεις και μέτρα που κανονικά θα εξασφάλιζαν το ότι ε, δεν δημιουργείται αυτό το απόθαμα προστασίας ε, μέσω ανακεφαλοποίησεως για να μειώσει τη μόχλευση που έχουν οι τράπεζες μέσω μειώσεως των πιστώσεων. Παρ' όλα αυτά, το πακέτο ανακεφαλοποίησεως σχεδιάστηκε από το ΕΚΟΦΗΝ σαν κομμάτι μεγαλύτερου πακέτου που αφορούσε κυρίως την βελτίωση της διακυβέρνησης αλλά ακόμα σημαντικότερο τμήμα είναι να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό τείχος για να μην μεταδίδεται η κρίση από ένα κράτος σε άλλο, η κρίση του κρατικού χρέους. Δυστυχώς, παρόλο που η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ ήταν ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα πακέτο, Τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι τα μέτρα ανακεφαλοποίησης που ανακοινώθηκαν και εισήχθησαν μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ήδη εφαρμόστηκαν όταν το τείχος προστασίας έχει οικοδομηθεί μόνο κατά το ίμιση για να το πω ήπια. Αυτό δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα. Και μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Αν το επιθυμεί η Επιτροπή βέβαια. Και τέλος, βέβαια συμβάλαμε στην προετοιμασία καθοδόν προς το Συμβούλιο της 9 Δεκεμβρίου. Στόχος της Προεδρίας ήταν η συνθήκη που θα ήταν αποτέλεσμα του Συμβουλίου να είναι συνθήκη των 27. και να εδράζεται επί κοινοτικής προσεγγίσεως. Όπως γνωρίζετε δυστυχώς αυτό απεδείχθη ε, αδύνατον, κρίμα, πολύ κρίμα. Να, να πω και κάποια άλλα για τους στόχους μας παρόλο που λίγη Προεδρία. Να πω κάποια λόγια για τους στόχους μας. Τους στόχους της πολωνικής κυβέρνησης. Όσον αφορά τη διακυβερνητική συνθήκη. Πρώτα απ' όλα. Κάτι πετύχαμε. Σημαντικό τμήμα αυτού είναι η ενίσχυση ε, του, ε, του Ταμείου του Νοσμονετικού Ταμείου, η γενική προσέγγιση που ακολουθήσαμε στον αφορά τις συνθήκες και δεν ζητώ συγγνώμη που δεν είπα αναφέρομαι στο θέμα, διότι είναι μια συνθήκη που αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και αφορά και το ΕΚΟΦΗΝ και την Επιτροπή σας. Η γενική προσέγγιση στη συνθήκη ποια ήταν. Ότι είμαστε υπέρ περαιτέρω εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση εντός Ευρωζώνης χωρίς να δημιουργηθούν νέες διαιρέσεις μεταξύ 17 και 10. Και πώς το βλέπουμε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό χρησιμοποιώντας εκτεταμένα τη συμμετοχή των ψήφων. Όλες οι χώρες να είναι παρούσες, με άλλα λόγια, όταν διεξάγονται οι συζητήσει για την Ευρωζώνη, αλλά να ψηφίζουν μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης. Διαφορετικά, περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωζώνης θα οδηγήσει σε περαιτέρω διέρεση μεταξύ των 17 και των 10. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται. στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της περαιτέρω, της εμβάθυνσης της Ευρωζώνης. Και αυτό αναπόφευκτα απαιτεί συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Κυρίως αν αυτή η εμβάθυνση προχωρούσε πολύ και απαιτούσε αυτό που συζητήθηκε, δηλαδή να επιστρέφονται οι προπολογισμοί πίσω στα τεχνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα μπορούσε να είναι αποκλειστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρέπει να πάρουμε μαθήματα την κρίση. είναι αρκετά σαφές ότι είναι μια κρίση μολυσματική θα έλεγα, απομόλυνση. Δεν είναι θέμα σφάλματος και λανθασμένης δημοσιονομικής πολιτικής. Πιστεύουμε συνεπώς ότι είτε χρειαζόμαστε σαφήνεια όσον αφορά το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση μόλυνση και διάδοση του φαινομένου και αν δεν υπάρχει σαφήνεια στι τρέχουσε ε, συνθήκες τίποτα δεν θα εμπόδιζε νομίζουμε να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αυτόν τον τρόπο βάσει των ισχυουσών συνθήκων. Αλλά αν δεν μπορεί να κινηθεί για να σταματήσει τη διάδοση του φαινομένου η ΕΚΤ στο πλαίσιο ε, τη ισχύουσα συνθήκη να αλλάξει εντολή που τη δόθηκε. Να τις επιτρέψει ε, να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και να δράσει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακαιρεότητα, αν θέλετε, ε, της ε, Ευρωζώνης ή ακόμα και η φερεγγιότητα κάποιου κράτους μέλους απειλείται από διάδοση του φαινομένου. Ζητώ συγγνώμη αν δεν ανέφερα κάποια άλλα σημαντικά πράγματα που έγιναν κατά έκα της Προεδρίας μας. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ομόλογα σταθερότητας, η ετήσια έκθεση ανάπτυξης, η μεγάλη μεταρρύθμιση ρυθμιστική που κάναμε, η συζήτηση του ενεργειακού φόρου, συζήτηση για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, συζήτηση για την ενοποίηση της φορολογικής βάσης για την φορολόγηση των εταιριών έγινε. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή η συζήτηση που διεξήχθη, αλλά επικεντρώθηκε επί των ζωτικότερων στοιχείων και των σημαντικότερων ε, του τελευταίου εξαμήνου. Θα έκλεινα λέγοντας ότι το Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου, όπως το βλέπω προσωπικά, με έδειξε τις πρώτες, ε, τα πρώτα ίχνη για κάποιο φως στο τέλος της σύραγγας. Μετά από 1,5 χρόνο ακολουθώντας λάθος κατεύθυνση, τελικά αρχίζουμε να κινούμαστε προς σωστή ενθαρρύνομαι πολύ από την απόφαση αυξήσεως των πόρων που θα διατίθεται προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διάφορες αποφάσεις για ενίσχυση του FSF και του ESM. κάπως καλυτερεύουν τα πράγματα. Ελήφθησαν πολύ χρήσιμες αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εβδομάδα που προηγήθηκε τη Συνόδου Κορυφής. Η κυρία Πρόεδρος θα αποφασίσει τι θα κάνουμε τώρα στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι όντω έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο σε πολλά ζητήματα επί Πολωνική Προεδρία. Το short selling και τα CDS, μάλλον τα ολοκληρώσαμε σχεδόν, όχι πλήρω. Και πολλά έγιναν στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ε, αναφέρατε τα επιτόκια τα οποία μπορεί να είναι τιμωρητικά για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα ανάκαμψης. Και ήδη το είδαμε από την αρχή της χρονιάς, καθυστερήσαμε πολύ και το όλο ζήτημα κόντεψε να επηρεάσει και άλλα μέλη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η βιωσιμότητα που επιδιώξαμε μας έφερε σχετικώς ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, να σας πω ότι το απόγευμα θα συζητήσουμε ξανά στην Επιτροπή των κανονισμό ΣΕΠΑΡΤ. Ε, μας έχουν πει ότι έρχεται από την Κορεπέρ, ε, είναι στο δρόμο το, η όλη πρόταση. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι επίσης μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσουμε Πολωνικής Προεδρίας. Και αναγνωρίζουμε ότι παρά τους κλειδονισμούς που προκάλεσε η κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εξετάζει εντελεχώς ζητήματα που αφορούν την ενιαία αγορά, τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και το πρωταρχικό ζήτημα του ευρώ. Ε, η συμφωνία ήταν κάτι σαν ψήφο εμπιστοσύνη προς το ευρώ. Αυτό ούτω ή άλλω είναι καθοριστικό για το γενικότερο έργο μα και ελπίζω ότι θετικά θα είναι τα αποτελέσματα και για του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Τώρα να περάσουμε στι παρεμβάσει των μελών. Πρώτο, ο Ζαν Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, να διαπιστώσω ότι η Πολωνική Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά. Τη προάλλε στην Ολομέλεια, παρουσία του Πρωθυπουργού σα, πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που τόνισαν ότι ήταν μια από τι καλύτερε προεδρίε που έχουμε γνωρίσει. Πραγματικά, σε καιρού θυελώδες, χρειάστηκε να πάρετε το τιμόνι για χάρη στη δουλειά σα σε όλους τους υπεύθυνους της Προεδρίας σας καταλήξαμε σε θετικά αποτελέσματα. Το θύμισε η Πρόεδρος. Το νομοθετικό κυνήγι, το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλάβατε να φέρετε εις πέρας ήταν φορτωμένο. Ήταν δύσκολη καιρή. Κι όμως ε, επιζήσατε αυτούς τους έξι μήνες Θυμήσατε προηγουμένω ότι εγκρίναμε το πακέτο τη διακυβέρνηση. Δύο κείμενα είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμπληρωθεί. Το πακέτο αυτό φαίνεται ω ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο τη οικονομική ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χωρών. Όμω βλέπουμε ότι από τη στιγμή που εγκρίθηκε, αμέσω μετά αρχίζουν να συζητούν τη διακυβερνητική συνθήκη τα κράτη-μέλη για την οικονομική διακυβέρνηση. Κάτι που στο Κοινοβούλιο είχε συζητηθεί πριν από ένα οκτάμινο και φαινόταν τότε τελείω ανέφικτο. Εσεί που ζήσατε μέσω αυτών των ε, συγκρούσεων. Μπορείτε να μας πείτε εάν παραμονές Χριστουγέννων μπορούμε να αποστείλουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα όπως αυτό που μας αναφέρατε. Δηλαδή υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Η φάτνη θα φωτιστεί Θυμίζω και την ωραία πολεμική βραδιά που μας οργανώσατε τις προάλλε από την πλευρά της Προεδρίας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι έχετε να πείτε εσεί για αυτό το θέμα που φαίνεται πολύ παράλογο για του συμπολίτε μα. Από τη μια ανακοινώνουμε ότι βρέθηκε κοινοτικό μέτρο για να ευνοήσουμε την οικονομική ολοκλήρωση και την άλλη πρέπει τα κράτη να σχεδιάσουν νέα συνθήκη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τη διαδικασία κυρωσή τη. Και θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Ξέρετε ότι την προηγούμενη άνοιξη με την προηγούμενη Προεδρία ε, ε, ζητήσαμε μια πολύ μικρή τροποποίηση του άρθρου 136 τη συνθήκη και ω σήμερα κανένα από τα κρατημέλη δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωση τη τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλά Χριστούγεννα. Monsieur Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. δεν θα μπορούσα εγώ και δεν ξέρω και πώς να το κάνω να προασπιστώ τα άλλα κράτη και ιδίως στην Πολωνία. Νομίζω η μόνη δυνατή εξήγηση είναι και εύλογη. Δηλαδή, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου η κατάσταση στην Ευρωζώνη, η ε, κατάσταση στο πλαίσιο αυτής της κρίσης του κρατικών χρεών δεν βελτιώθηκε δεν βελτιώθηκε. Φυσικό είναι τα κράτη να προσπαθούν να επιστρέψουν σε ιδέες που δεν είχαν γίνει αποδεκτές προηγουμένως. Γιατί κάποια από τα σημαντικότερα κράτη, ιδρυτές της Ένωσης, δεν τις δέχονταν. Θα Συνέχιζα ίσως τα αγγλικά, θα έλεγα μάλλον στα αγγλικά, καλύτερα καλή αργά παρά ποτέ. Νομίζω τα προβλήματα που διαβλέπετε για την κύρωση δεν θα είναι αυτά που θα δημιουργήσουν το πρόβλημα, που θα εμποδίσουν την ε, κύρωση. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Uh, next, I have ο Βέρνερ Λάγκεν ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Μια στιγμή. Ja, suche noch die Sprache. Eins. Κανάλι 1. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και όλες τις υπηρεσίες σας για την πάρα πολύ εντατική εργασία που έκανε για διάφορα συγκεκριμένα νομοθετήματα και το ανέφερε ήδη η πρόεδρος μας. Εγώ υπήρξα εισηγητής για τα ε, παράγωγα over the counter, τα εκτός αγοράς και εμείς από ό,τι είδαμε λοιπόν δεν ήταν ο στόχος μας να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε λύσεις για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται και οι θεσμικές υποχρεώσεις σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Λέει η συνθήκη ότι οι αποφάσεις παίρνονται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο να αποφασίσουν με ειδική πλειοψηφία. Επομένως και στη δική σας περίπτωση του Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει λήψη απόφαση με ειδική πλειοψηφία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι υπάλληλοι τη Πολενική προεδρίας λειτουργήσαν πολύ καλά, δεν κατάφερε το ΕΚΟΦΗΝ να καταλήξει σε συγκεκριμένες λύσεις σε ορισμένα θέματα γιατί ζήτησε να γίνονται οι αποφάσεις με ομόφωνο τρόπο και όχι με ειδική πλειοψηφία όπως προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Βλέπω ότι όλο και λιγότερο και φαινόταν αυτό και στην Ουγγρική Προεδρία. Όλο λιγότερο χρησιμοποιείται η φυσιολογική διαδικασία νομοθεσίας βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να το διαπιστώσω αυτό. Το είδα αυτό για, τις εκτός αγοράς, για τα εκτό αγοράς παράγωγα. Στο τέλος της διαδικασίας το ΕΚΟΦΗΝ δεν μπορούσε να καταλήξει σε μια λογική λύση σε σχέση με τις εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχέσεις με τρίτες χώρες να βρει. Αυτό δεν οφείλεται στου ειδικού σα υπαλλήλου. Και στην Κορεπέρ πρόκειται για το γεγονό ότι το ΕΚΟΦΗΝ μπλοκάρισε την απόφαση. Σα λέω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να δεχτεί αυτό ότι υπάρχει μια μόνιμη παράκαμψη της συνθήκης Λισαβόνας. Δεν πρόκειται για σας, πρόκειται για όλους τους Υπουργούς Οικονομικών. Έχετε εδώ παρουσιάσει ένα απολογισμό. Σίγουρα είχατε αναλάβει ευθύνε σε ένα πολύ δύσκολο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά για την ε, αλλαγή της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είπατε τίποτα. Και επίσης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Βλέπουμε να υπάρχει ακόμα η διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας 3 και μέχρι το 2018 θα πρέπει να φτάσουν 10% το ίδιο κεφάλαιο οι τράπεζες. Το stress test έγινε με 9% ίδιο κεφάλαιο και με μία διαφορετική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων. Πώς μπορείτε λοιπόν να καταλήξετε σε μια σαφή γραμμή όταν έχετε διαφορετικές και πολλές φορές αντιφατικές αντιμετωπίσεις στα stress και στη Βασιλεία 3. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση των G20 ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς να υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία. Εσείς δεν έχετε πει τίποτα για ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων και φορέων. Εγώ λοιπόν είμαι πραγματικά απογοητευμένος από τα αποτελέσματα ενώ πρέπει να επενέσω τη διαδικασία που ακολουθήσατε και τη λειτουργία σα ω Προεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο των συνεργατών μου θέλω να σα ευχαριστήσω για το θέμα τώρα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Συμβούλιο Κοφίν και του τρόπου λήψη αποφάσεων. Θέλω να το πω αυτό πολύ σαφώς. Το γεγονός ότι το ΕΚΟΦΗΝ μπορεί να πάρει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Και πιστεύω ότι θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την άποψη, τουλάχιστον αυτή είναι και η λογική που ακολουθεί κάθε Προεδρία, αποφασίζει πώς θα δράσει. Και εγώ θα παραμείνω πιστός σε αυτή την άποψη, όχι μονάχος Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοφίν αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Και θα ήθελα αυτό να γίνει σαφές. Για την εφαρμογή της Βασιλείας 3 και το 9% κεφάλαιο πυρήνος. Στάθμης 1, δηλαδή τύρα 1. Εδώ νομίζω ότι υπήρξε ο φόβος ότι αν υπάρχει ανεπαρκές κεφάλαιο των τραπεζών στις τωρινές συγκυρίες, ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πάγωμα, σε ένα στέγνομα της διατραπεζικής αγοράς. Αυτός είναι ο φόβος, δεν σας λέω την πραγματικότητα. Η ταχεία αντίδραση η οποία κατά την άποψή μας θα εξασφάλιζε στην αγορά ότι όλες οι τράπεζες θα έχουν την απαραίτητη κεφαλαιοχική επάρκεια μέχρι τα μέσα του 2012, αυτό θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να αποτρέψει μια σοβαρή ύφεση η οποία θα μπορούσε να προκύψει από το στέγνομα της διατραπεζικής αγοράς. Δυστυχώς. Και όπως και η Πολωνία ως Προεδρία και όπως άλλες χώρες συμφώνησαν, η γενική άποψη του Συμβουλίου Ακοφίν ήταν ότι θα ήταν σφάλμα να προχωρήσουμε με το πακέτο επανακεφαλαιοποίησης, χωρίς προηγουμένως να έχουμε το τείχος ασφαλείας, το firewall δηλαδή, γιατί φοβόμασταν ότι μπορούσε να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, βάσει του οποίου η επανακεφαλαιοποίηση θα επέβαλε περαιτέρω άχθος στο, στα κρατικά ομόλογα, θα μειωνόταν η αξιολόγησή τους και αυτό θα επέβαλε περαιτέρω βάρη, βάρος στις τράπεζες. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα σφάλμα και το έχει τονίσει ο Μάριο Ντράγκη σε πολλές ευκαιρίες. Το είπε και χθε και νομίζω ότι συμφωνώ μαζί του. Θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει το τείχος ασφαλείας, το firewall. Ακολουθήσαμε τη λαθασμένη πορεία λοιπόν, τη λαθασμένη σειρά. Τώρα προχωρούμε <clears throat> με το τείχος ασφαλείας αλλά δεν έχει νόημα να παριστάνουμε ότι δεν κάναμε λάθο όταν έχουμε κάνει λάθο και είναι καλύτερο να το παραδεχτούμε δημόσια και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση από αυτό το σημείο και πέρα. Και να προσπαθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να επανορθώσουμε. Για τα άλλα θέματα που θίξατε, εγώ σας ζητώ συγγνώμη αν κάποιος θεωρεί ότι εγώ δεν κατάφερα να αναφέρω σημαντικά ζητήματα και αυτά που είπατε είναι σημαντικά ζητήματα. Συμφωνούμε απόλυτα με τα συμπεράσματα των G20 και την εντολή τους για την ε, εποπτεία και τη ρύθμιση όλων των εμπλεκομένων ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Εγώ θέλησα να παραμείνω πιστό στον χρόνο που μου έδωσε η πρόεδρος, η κυρία πρόεδρος και γι' αυτό ίσως παρέλειψα ορισμένα σημεία και προχώρησα ορισμένα θέματα, σε ορισμένα θέματα πολύ γρήγορα. Ο επόμενος ο μιλητή είναι και η Σουίνμπερν. Ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε στις στη σας να μιλήσετε και πρέπει να σας συγχαρούμε και ως εκπρόσωπος του ECR θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριλάβατε όλους τις συζητήσει και όπως κινηθήκατε σαν Πολωνική Προεδρία και πρέπει πολλές ώρες ε, να συμμετέχω σε τριμερείς ε, διαλόγους ε, για το six pack και για άλλα θέματα και πάντα με επαγγελματικό τρόπο οργανώσατε συζητήσεις και αυτό δείχνει πόσο ισχυρός ηγέτης ήσασταν και οι άλλοι. Πρέπει να πω ότι έγιναν ανταλλαγές απόψεων ε, και εδώ στην Επιτροπή σχετικά με το πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ευρώπη ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι έτοιμοι τελικά να δώσουν χρήματα και να μην δίνουν μόνο υποσχέσεις καταφέρατε να μου εξηγήσετε το θέμα αυτό και να με κάνετε να πιστέψω ότι πραγματικά καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει η σωστή επικοινωνία με τις αγορές. Τι συμβουλή θα δίνατε στην επερχόμενη Προεδρία της Δανίας, πώς θα μπορούσε να βελτιώσει την επικοινωνία με τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, ώστε να καταφέρει να αποκαταστήσει κάποια εμπιστοσύνη στους επενδυτές ότι η Ευρώπη είναι ένα καλό σημείο να κάνει κανείς επενδύσεις και με σχετικά χαμηλό κίνδυνο συγκρίση με άλλα σημεία του κόσμου. Απάντηση. Έχω την εντύπωση ότι η επικείμενη ε, Δανέζικη Προεδρία θα συμπεριλαμβάνει όλους την προσπάθεια. Σίγουρα θα σεβαστεί πλήρως το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό, όπως και εμείς, ως Πολωνική Προεδρία. Όσον αφορά την ε, επικοινωνία, ε, θα πω ξανά ότι ενό προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ έχει πολύ σημαντικές ε, δεξιότητες όσον αφορά την επικοινωνία και ένα στοιχείο που θα βοηθήσει την επικοινωνία, θα βοηθούσε την επικοινωνία και ελπίζω θα βοηθήσει την επικοινωνία, είναι και το εξής. Αν η νέα διακυβερνητική συνθήκη, δυστυχώς διακυβερνητική συνθήκη εξασφαλίζει συμμετοχή όλων των μελών του Euro, στο Eurogroup και στις συνεδριάσεις της Ευρωζώνης. Διότι έτσι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης και θα διευκολυνθεί στο έργο της η Προεδρία. Αν δεν είναι Προεδρία Ευρωζώνης, θα τη βοηθήσει να επικοινωνεί με λογικό τρόπο με την αγορά. Εμείς τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σαν Πολωνική Προεδρία στην επικοινωνία με τις αγορές ήταν ότι κάποιες φορές δεν γνωρίζαμε όχι τι αποφασιζόταν στις ε, ομάδες της Ευρωζώνης, αλλά ποια ήταν η μορφή της συζήτησης, το πνεύμα της συζήτησης. Και ήταν δύσκολο τελικά να παρουσιαστεί μια ομοιόμορφη εικόνα σε όλους τους θεσμούς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωζώνη, Eurogroup. θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον τα προβλήματα σε επίπεδο των διαφόρων χωρών και αν υπάρχει ουσία θα υπάρχει και επικοινωνία. Αυτό το ένα συνεπάγει το άλλο. Αν δεν υπάρχει ουσία, τι να σου κάνει η επικοινωνία. αυτό έχω να πω και ευχαριστώ. Όσον αφορά τώρα αν έχουμε ουσία και επικοινωνία, αν έχουμε ουσία, η Δανέζικη Προεδρία θα μπορέσει να την προβάλλει εξαιρετικά καλά. Και κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Είπα προηγουμένω ότι αρχίσαμε την οικοδόμηση του τείχους προστασίας, του firewall. Ε, έχουμε προβλήματα με την ολοκλήρωση του τείχους. Πρέπει να δούμε το πώς οι πρόσφατες αποφάσεις κυρίως αυτή που αφορά την ε, μακροχρόνια ρευστότητα που θα χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τις τράπεζες, κατά πόσο αυτό θα είναι κάτι ε, επιτυχές και σταθεροποιητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω τον υπόλοιπο κατάλογο. Καταρτίστηκε από τη Γραμματεία ανάλογα με το πώ προσήλκει ο καθένα την προσοχή τη γραμματεία, ίσω να μην σωστή σειρά. Λίζα Φεραίρο, Όλε Σμιτ. Αυτοί είναι οι ομιλητέ. Άλλο που θέλει να μπει στον κατάλογο των ομιλητών. Καλώ. Λίσα. Well, thank you very much and thank you for being... ε, ευχαριστώ και ευχαριστούμε που ήρθατε. Νομίζω σκοπό τη σημερινή συζήτηση δεν είναι απλώ να εκφράσουμε τι ευχαριστίε σα για το έργο, για το έργο σα. Γιατί ούτω ή άλλω σα ευχαριστούμε ειλικρινώ για τον ορθολογικό τρόπο που ασχοληθήκατε με τα τιμωρητικά επιτόκια για τη δουλειά σα στο Sixpack όπου υπήρξε εισηγήτρια μία των εισηγητών. Σας Ευχαριστούμε λοιπόν για όλο αυτό το έργο, αλλά νομίζω σε αυτήν την στιγμή μπορείτε να αισθανθείτε απελευθέρωση. Και ήθελα και εγώ να αξιοποιήσω αυτό το συνέστημα ώστε τη σύστασή σας να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα αυτό και στο ερχόμενο εξάμεινο να την ε, ακολουθήσουμε, να την αξιοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί. Ένα από τα προβλήματα που νομίζω ότι παραμένουν είναι ο συσχετισμό και ο φαύλο κύκλο που δημιουργήθηκε μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα και των τραπεζών που κλειδονίζονται. Αυτό δεν έχει πάψει. Νομίζω οι ιδιωτικέ δεσμεύσει στο ζήτημα του κρατικού χρέου ήταν ένα από τα σφάλματα κατά τη δική μου άποψη που έγιναν κατά την πορεία. Όμω το να Επιζητούμε λύσει στα δύο αυτά ζητήματα. Είναι σημαντικό. Πόσο πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε μακριά για να αντιμετωπίσουμε τις χώρε που κινδυνεύουν. Το μοντέλο που ξεκίνησε να αναπτύσσεται δεν πρέπει να συμπληρωθεί. Ασχοληθήκατε με το SM, το IMF, το EFSF στην θητεία σας. Θεωρείτε ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα λειτουργήσουν και πώς. Πιστεύετε ότι όσα πετύχαμε στο Six-Pack συμπεριλαμβανόμενης της μακροοικονομικής εποπτείας αντικατοπτρίζονται επαρκώς στο κείμενο που ξέρουμε ότι πρόκειται να προταθεί μέσω της προσέγγισης ε, και της διακυβερνητικής συνθήκης για την οικονομική διακυβέρνηση και για τις τράπεζες. Δεν πιστεύετε ότι ένας από τους κρίκους που λείπει είναι μια δομή για την αντιμετώπιση των κρίσεων σε ό,τι αφορά τι τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή μα είπε ότι το επεξεργάζεται το θέμα, αλλά επιφυλάσσεται για να διστάζει να υποβάλει κάποια πρόταση. Δεν νομίζετε ότι για να αντιμετωπιστούν τέτοιε κρίσει από τι τράπεζε θα χρειάζεται μια συγκεκριμένη δομή. Τον ζήσαμε τον φαύλο κύκλο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά ζητήματα, πιστεύω, με έναν τρόπο συνεπή. Σας ευχαριστώ. Για να περάσουμε απευθείας στην ουσία του ζητήματος, εφόσον ρωτάτε. Πολλά μπορεί κανείς να επιτρέψει στον εαυτό του να κάνει, αν έχει απαραίτητα προστατευτικά. Ε, εάν υπήρχε αυτό, αυτή η πρόνοια, δεν θα, χρειαζόταν, δεν θα ήταν πρόβλημα το PSI, όπως και η επανακεφαλοποίηση των τραπεζών με τα σχετικά μέτρα. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν είχαμε προστατευτικά συστήματα και δομές. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να υπάρχει απαραίτητη πρόνοια, τα προστατευτικά μέτρα. και όσο ότου ως αποκτήσουμε τέτοια δίχτυα ασφαλείας, πείτε το όπως θέλετε, προστατευτικούς μηχανισμούς, τέλος πάντων δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος για το τι θα μπορεί να κάνει με ασφάλεια στην μετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένω να αναδυθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διαχείριση τη Παρόλο που θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα ή ένα πλαίσιο για την επίλυση των ε, τέτοιων ζητημάτων, ώστε να μπορούν οι εθνικέ κυβερνήσει να εισαγάγουν κάθε φορά στην εθνική του νομοθεσία τι απαιτούμενε διατάξει. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα κενά που παραμένουν στο πλουστάσιο μας, διότι όλοι έπρεπε να προχωρήσουν και να βρουν λύσεις ad hoc, ανάλογα με τις περιστάσεις που παρουσιάζονταν. Το οποίο ίσως είναι και καλύτερο, γιατί δεν ήταν δυνατόν όλα να είναι ετοιμασμένα και όμορφα σχεδιασμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απλώς μετά να ξεπατικώνονται. Θα ήταν ακόμα καλύτερα βέβαια αν εάν υπήρχε μια προσέγγιση ενιαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως και ταχύτερη η πορεία μας. Αλλά είναι δυσεπίλητα τα ζητήματα αυτά. Τώρα για την συνθήκη έναντι του ΣΥΚΣΠΑΚ. Νομίζω ότι ο κύριο Λάγκεν το είπε προηγουμένως. Η συνθήκη σε μεγάλο βαθμό ήταν η αρχικό σχεδιασμός που είχαμε κατά νου για το ΣΥΚΣΠΑΚ. Όμως Είναι καλό να διδάσκεται κανείς από τα σφάλματα που έχει διαπράξει. Ναι, δίκιο είχατε. Δεν έχω καμία δυσκολία να το παραδεχτώ. Θα σας το πω ειλικρινώς. Το κοινοβούλιο είχε δίκιο. Τουλάχιστον έχουμε ευτυχώς το περιθώριο να διορθώσουμε τα σφάλματά μας είναι καλύτερο από το να λέμε ότι εφόσον κάναμε ένα λάθος θα συνεχίσουμε στη λανθασμένη πορεία στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Κάποια πράγματα λειτουργούν, κάποια όχι. Πριν δώσω το λόγο στο επόμενο μιλητή, ήθελα να πω ότι ορισμένε από τι πρόνοιε οι οποίε εφαρμόστηκαν, όπω τα συστήματα παροχή ρευστότητο της Κεντρικής Τράπεζας είναι σημαντικά γιατί μειώθηκαν τα ισπανικά επιτόκια σε σημαντικό βαθμό χάρη στις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας. Ο Όλες συμμετέχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου αρέσει το ύφο με το οποίο μιλάτε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά η Πολωνική Προεδρία αφήσατε τα εσωτερικά σας θέματα έξω από το Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα, παρά το γεγονός ότι ήταν προεκλογική περίοδος στις, ε, στη χώρα σας και το εκτιμώ αυτό. Έχετε δείξει μεγάλη αισιοδοξία. Εγώ είμαι φιλελεύθερος και εγώ είμαι κανονικά αισιόδοξο. Βλέπετε κάποιο φως στο τέλος του τούνελ που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα το φως αυτό. γιατί βλέπω επίσης και τα πρώτα βήματα στο διχασμό της Ευρώπης. Κάποιοι από εμά μένουν απ' έξω. Έρχομαι από μια μικρή χώρα στη Βόρεια Ευρώπη και ανησυχούμε τα μάλα. <clears throat> Ελπίζουμε, και το είπατε και εσείς ο ίδιος, ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούμε εκτός του νυμφόντος ή δεν θα βρεθούμε σε κάποια φάση που δεν θα μπαίνουμε καν στην αίθουσα όταν συζητάμε οικονομικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε πώς θα μπορούσαμε να ξαναέρθουμε σε μια αντιμετώπιση από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει 27 ή 28 ίσα μέλη. Κάνατε και μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ιστορικού χαρακτήρα για κάποιους από τους γείτονές σας. Και αυτό ήταν κάτι που σχολιαστήκε στη δική μου χώρα. Ο φόβος μας λοιπόν είναι ότι δεν θέλουμε να μας διαχειρίζονται οι μεγάλες χώρες στην Ευρώπη. <clears throat> Αλλά ο φόβος είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει το πάνω χέρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέσει η Γερμανία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Πρέπει να πουλήσουμε και τα προϊόντα μας στα αυτούς. Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί μια ένωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να πω ερχόμενος από μια μικρή χώρα και είχαμε την ίδια συζήτηση και με τους Δανούς. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα θέματα αυτά και ελπίζω ότι θα μπορούσατε να πείσετε τους συναδέλφους σας ότι οποιαδήποτε μορφή καταμερισμού της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες, σε διαφορετικά στρατόπεδα είναι κάτι το αντιπαραγωγικό και κάτι το επικίνδυνο ξέρουμε και εμείς την ιστορία της Ευρώπης και εσείς, εσείς θα την ξέρετε πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι θεωρούμε ότι μια διαίρεση της Ευρώπης σε οποιαδήποτε στιγμή χρονική, αλλά ιδίω τώρα θα ήταν μια πλήρης καταστροφή, μια με τεράστια καταστροφή. Αλλά παράλληλα είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε διάσπαση της Ευρωζώνης θα ήταν εξίσου ολέθρια. Γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο αυτό και τον μιλώ με, ως Πολωνός αλλά αυτό είναι και το πνεύμα το οποίο διέπει την Προεδρία μας και γι' αυτό νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να μιλήσω έτσι σήμερα θεωρήσαμε ότι η μόνη λογική απάντηση στα προβλήματα αυτά ήταν να υποστηρίξουμε πλήρως την βαθύτερη ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη, ενώ συγχρόνως τονίζαμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η βαθύτερη ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαχωριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωζώνη και σε αυτούς που είναι εκτός της Ευρωζώνης και ο μηχανισμός που μπορεί να μας εξασφαλίσει να το πετύχουμε αυτό είναι ακριβώς <clears throat> ο μηχανισμός αυτός συμμετοχής αλλά όχι Λήψη συμμετοχής στη λήψη απόφαση, δηλαδή όχι δικαίωμα ψήφου, που προβλέπεται για την ενισχυμένη συνεργασία από τις συνθήκες. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τον δρόμο αυτό, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε τις χώρες της Ευρωζώνης προς την κατεύθυνση της βαθύτερης ολοκλήρωσης που θέλουν να επιτύχουν, χωρίς συγχρόνως να διακυβεύεται και η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου και είναι κατά κάποιο τρόπο ευτύχημα ότι η Προεδρία βρέθηκε στα χέρια μιας χώρας που δεν ήταν στη ζώνη του ευρώ <clears throat> καταρχήν της Ουγγαρίας, μετά στα δικά μας χέρια και μετά της Δανίας που και αυτή δεν βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ. Για το θέμα των μεγάλων κρατών και της ε, υπεροχής, του τους δεν ήταν αυτά που είπα εγώ, τα είπε ο υπουργό Εξωτερικό μας, ο κ. Σικόσκι. Αυτός είπε ότι ανησυχούσε περισσότερο για την αδράνεια της Γερμανίας από ότι για την επιβολή της θέσης της Γερμανίας. Αυτό οδήγησε και σε κάποιες εκπλήξεις και κάποια εμβροντισία, αλλά πράγματι η άποψή μα είναι έτσι και λόγω και τη γεωγραφική μα θέση. ότι πιστεύουμε ότι η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό θέμα για μας, είναι και ένα θέμα εθνικής ασφάλειας για μας, τους Πολωνούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μαρία Τάισεν. Θα μιλήσω Ολλανδικά, Πρόεδρε. Ik wil me heel graag aansluiten bij de Με τα χαράς εγκρίνω τα επενετικά λόγια που απευθύνθηκαν προς την Πολωνική Προεδρία έκανε πολλή δουλειά επεκράτησε και καλή ατμόσφαιρα παρά τις δύσκολες συνθήκες ε, θέλω να αναφέρω ένα-δύο πράγματα απευθυνόμενοι προς τον Προεδρεύοντα όταν μιλήσατε για την ΕΚΤ είπατε ότι υπό κάποιες ε, περιστάσεις αν ο κίνδυνος μόλυνσης διάδοση του φαινομένου είναι πολύ μεγάλος και η κεραιότητα της Ευρωζώνης ε, απειληθεί ότι η ΕΚΤ θα έπρεπε να μπορεί να κινηθεί και να αλλάξει η συνθήκη αν τη επιτρέψει να κάνει περισσότερα. Ίσως πολλοί να συμφωνούν μαζί σας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της κρίσης, από τη στιγμή που θα επιστρέψει η πειθαρχία στα κράτη-μέλη, ότι αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει και τότε να εφαρμόζεται. Δεύτερον, η νέα διακυβερνητική συνθήκη που έχει προταθεί έχει συζητηθεί ήδη εκτενώ. Είδαμε χτε ένα κείμενο. Δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώ του εγγράφου που είδα. Διερωτώ με, αν πρόκειται να επεξεργαστούμε μια διακυβερνητική μέθοδο και απομακρυνθούμε από τη Λισαβόνα, ποιος είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του κειμένου, ποιος φέρει την ευθύνη λοιπόν. Μετά, με μια διακυβερνητική συνθήκη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ολοκλήρωση και μάλιστα με έναν τρόπο που να παραμένει νόμιμος από πλευράς δημοκρατικής. Διότι φαντάζομαι ότι αν πολλές αρμοδιότητες εκχωρηθούν από τα κάτι μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ε, δημιουργούνται μεγάλες ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινείται δημοκρατικά, να υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα για την εφαρμογή των νέων ε, κανόνων. Και διαβάζοντας το πρώτο κείμενο, έχω κάποια ερωτηματικά που μου δημιουργήθηκαν όσον αφορά αυτό το θέμα. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. I have some sympathy with what Καταλαβαίνω αυτά που λέτε κάπως. Καταρχήν δημιουργήσαμε θεσμούς ή σύστημα διακυβέρνησης που θα έπρεπε από τη στιγμή που θα βγούμε από την παρούσα κατάσταση εξασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό το φαινόμενο. Απ' την άλλη, η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να κρατήσει αρκετά. Η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι θα είναι θέμα ετών και όχι μηνών. Προσωπικά πιστεύω ότι το παρόν πλαίσιο της συνθήκης ε, επιτρέπει στην τράπεζα, την Κεντροπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει όσα προανέφερα. Όμως, ε, επειδή κάποιοι ερμηνεύουν τη συνθήκη με έναν τρόπο που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, θα είναι καλό να είναι σαφέ ότι επιτρέπεται να κινηθεί η πιο ελεύθερη τράπεζα. Και αν συνεχιστεί το φαινόμενο επί σειρά ετών, όπω δυστυχώ έτσι φαίνεται, τότε είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να γίνει. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αν βγούμε από την κρίση πολύ γρήγορα και μπούμε στο, στη διακυβερνητική συνθήκη και εντό του πλαισίου του Six Pack ίσως να είναι λιγότερο επίγον αυτό, αλλά πάντα βρήθη εκπλήξεων η ζωή. Τι να πω, άρα σοφόν θα ήταν εφόσον μας είπαν ότι αυτό που φαίνεται προφανώς σωστό στην τεράστια πλειοψηφία ε, των ε, οικονομολόγων αντιβαίνει τις συνθήκες. Εν τη αυτή περιπτώσει θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες όσον αφορά ε, τη συνθήκη αυτή καθ' Από ό,τι κατάλαβα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Βον Ρομπάι, συνέταξε το κείμενο και εκπρόσωποι των κρατών μελών θα αρχίσουν να το επεξεργάζουν το κείμενο σήμερα το απόγευμα. Για το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Εάν υπάρξει μηχανισμός πειθαρχίας για τα κράτη της Ευρωζώνης θα μπορούσε να είναι αυτόματος, ξεκάθαρα αυτόματος μηχανισμός από τη μια που εμπεριέχει αυτό προβλήματα διότι οι κανόνες δεν μπορούν κάθε κατάσταση είτε από την άλλη πλευρά αν υπάρχει διακριτική ευχέρεια εφαρμογής τότε η αρμοδιότητα θα πρέπει να δοθεί σε κάποιο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, εν τη αυτή περίπτωση, ισχύει αυτό που είπα στην αρχή. Θα απαιτείται σημαντικό επίπεδο δημοκρατικής νομιμότητας. Δηλαδή συμφωνώ με αυτό που μου είπατε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πού είναι ο κατάλογος των ομιλητών. Ο Σβέν έπρεπε να φύγει. Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να αναγνωρίσω το θετικό πνεύμα και την καλή πίστη που έχει δείξει η Πολωνική Προεδρία. Το γεγονός ότι θέλησε να είναι περιεκτική, να συμπεριλάβει όλους και φυσικά αν τα μοναχά τη θέλησή τη θα είχε πετύχει πολύ περισσότερα η Πολωνική Προεδρία. Έχουμε μια κρίση κρατικού χρέους, μια κρίση συγχρόνους και ιδιωτικού χρέους και έχει τεθεί και σε κρίση και το ίδιο το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κρίση, αν θέλετε, βιωσιμότητας. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε περισσότερο για το τι παραμένει ακόμα να γίνει. Δηλαδή τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και τι χρειάζεται να κάνουμε στο μέλλον. Κατά την άποψή μου υπήρξε ένα πρόβλημα διαχείρισης όταν φτάσαμε να έχουμε πολύ ψηλά επιτόκια διορθώθηκε αυτό υπήρξε πρόβλημα να αντιμετωπιστεί η επιμόλυνση, ε, υπήρξε πρόβλημα με την συμμετοχή των ιδιωτών που περιορίστηκε μονάχα στην περίπτωση της Ελλάδος, <clears throat> υπήρξε πρόβλημα και με την ανακεφαλαίωση όταν χρησιμοποιήθηκε το απλώς η τιμή αγοράς των ε, κρατικών ομολόγων και αυτό οδήγησε σε προβλήματα αβεβαίωτος. Υπάρχει τώρα το θέμα καταρχήν <clears throat> του κρατικού χρέους. Μιλάμε για λιτότητα σε δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά <clears throat> πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους με μια πολιτική ανάπτυξης, με μια πολιτική που θα τόνωσε την απασχόληση, ενδεχομένω με τα ευρωομόλογα. Ποια είναι η άποψή σα. Δεύτερον, το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Μήπως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εξηγηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να σκεφτούμε πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη στο να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία γιατί δεν έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα της ε, αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους στην περίπτωση του κρατικού χρέους. Σε ποιες παραμέτρους θα πρέπει να βασιστούμε για να κινηθούμε στο θέμα αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με τις συνθήκες. Όλες οι συνθήκες είναι διακυβερνητικού χαρακτήρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η τελευταία αυτή συμφωνία που έγινε μεταξύ 26 χωρών δεν είναι μονάχα διακυβερνητική, έχει και κάποιο ενωσιακό χαρακτήρα παρά τον διακυβερνητικό της χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο όμως να επιληθούν τα προβλήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια μεγαλύτερη αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει μεγαλύτερη ικανότητα δράση στο δημοσιονομικό τομέα, αλλά να έλκει την νομιμοποίησή της και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. για να ξεκινήσω με την τελευταία σας παρατήρηση. <clears throat> Εγώ πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι μια διακυβερνητική συμφωνία 26 χωρών σήμερα και 27 μετά από την ένταξη της Κροατίας δεν θα έβρισκε εύκολο να χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά εργαλεία, τα κοινοτικά θεσμικά εργαλεία. Κατανοώ λοιπόν <clears throat> τον στόχο σας από ό,τι κατανοώ εγώ θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χωρίς τη συνεργασία όλων των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση σε τιμές αγοράς του κρατικού χρέους. <clears throat> Αυτό ήταν ένα που σχεδόν κάναμε. Κάναμε ένα αντίθετο σφάλμα σχεδόν. Αν το κρατικό χρέος αποτιμήτωσε σε τιμή αγοράς, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε συνέχεια να επανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζες και αυτό θα αύξανε την ευθραυστότητα και το χρέος των ε, κρατών που θα μείωνε και την αξία των ομολόγων τους μέσα στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών. Αυτό είναι ακριβώς ένας φαύλος κύκλος. Γι' αυτό ήταν ουσιαστικό να έχουμε πρώτα ένα αξιόπιστο τείχος ασφαλείας ή θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό πρώτα για να μετριαστούν οι αρνητικές πτυχές της επανακεφαλαιοποίησης η οποία είχε θετικά στοιχεία αλλά έχει και αυτά τα το δυνητικά πολύ σημαντικό κίνδυνο της απομείωσης της αξίας των ομολογών. Κάναμε κάποια θετικά πράγματα μέσα στο πακέτο αυτό επανακεφαλαιοποίησης. Είπαμε ότι αυτή η διαδικασία αφορά <clears throat> ε, ε, τα κρατικά ομολόγα και την τιμή που είχαν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009 και είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν περαιτέρω μαξιλαράκια κεφαλαίου και να μην γίνουν αυτά από απομόχλευση εκτός στην περίπτωση που απλώς απεκδίεται μια τράπεζα ορισμένες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Και είπαμε πίσω ότι οι αρχές της Βιέννης για την παροχή ρευστότητα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τύχουν σεβασμού. Καταφέραμε με όλα αυτά να βελτιώσουμε την ποιότητα <clears throat> της επανακεφαλαιοποίησης της διαδικασίας αυτής. Το βασικό όμως σφάλμα ήταν ένα σφάλμα χρονισμού. Μόνο τώρα σιγά σιγά αρχίζει να επανορθώνεται. Ευτυχώς ο χρόνος περάτωσης της διαδικασίας επανακεφαλαιοποίησης που είναι το, τα μέσα του 2012 θα μας επιτρέψει να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία ενός αξιόπιστου τείχους ασφαλείας μέχρι τότε. Οπότε ο κίνδυνος του φαύλου κύκλου που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν κατάλαβα αυτά που είπατε για το ιδιωτικό χρέος. Ίσως μπορείτε να το επαναλάβετε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε για το ιδιωτικό τμήμα του χρέους. Εγώ θεωρώ ότι το ιδιωτικό χρέος, ότι ενώ για το δημόσιο χρέος υπήρξαν σαφές προδιαγραφές για δημοσιονομική λιτότητα, για το ιδιωτικό χρέος δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Απαιτείται λοιπόν αυτή η εξυγίανση μέσω της ανακεφαλαίωσης, ανακεφαλαιοποίησης, και θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό με ένα ευρωπαϊκό τρόπο, ποιος θα είναι και ο ρόλος του EFSF στην διαδικασία συμπλήρωσης αυτής της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Σύμφωνο, σύμφωνο μαζί σας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα από αυτά. Έχουμε τη διαδικασία για τις υπερβολικές ανισορροπίες στο Six που λαμβάνει υπόψη το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε το EFSF που διατίθεται στις χώρες της Ευρωζώνης. Έχουμε ένα Συμβούλιο Ανάλυσης Τιμικού Κινδύνου που εξετάζει ε, το ιδιωτικό χρέος σαν ενδεχόμενη πηγή μελλοντικής κρίσης. Τι να πω, συμφωνώ εν τη εννοία ότι πάντα μπορεί να καταφέρει κανεί καλύτερα, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημη η κατάσταση στον αφορά το ιδιωτικό χρέο. Εκτό από το γεγονό ότι ίσω. ίσως δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε το γεγονός ότι οι πραγματικές πηγές ανάπτυξης δεν βρίσκονται απαραίτητα στον όγκο πίστο σε σχέση με το ΑΕΠ. Οπότε έρχομαι στο πρώτο ερώτημα σα, Τι πρέπει να κάνουμε. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε θετικέ μεταρρυθμίσει που θα απελευθερώσουν τι αγορέ και πάνω απ' όλα τι αγορέ εργασία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Για να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη αυτή θα μας επιτρέψει ε, να περάσουμε το βουνό του δημοσίου χρέους που δημιουργήσαμε. Να το σκαρφαλώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σιλβί, είσαι επόμενη. Ίσως ε, δεν θα σε πειράζει να μιλήσει. Έχουμε χρόνο και άλλες ερωτήσει. Αν κάποιος άλλος θέλει να ξανακάνει ερώτηση, το χέρι θέλετε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, για... Ευχαριστούμε την Πολωνική Προεδρία για όλο αυτό το έργο. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε το σχέδιο συνθήκης όπως το πληροφορηθήκαμε. Γιατί εμένα μου προκαλεί έντονες ανησυχίες. Καλό θα ήταν να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό για τους εξή δύο λόγους. Αυτά συνδέονται άμεσα και με την Προεδρία σας. Πρώτον, το six διότι και εσείς ο ίδιος το είπατε, η συνθήκη αυτή αναλαμβάνει ένα μέρος από το six και το επαναλαμβάνει. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, ε, Είχαμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να μα δίνετε και απαραίτητη σημασία όταν βλέπουμε μία πτυχή ενό ιδιαίτερα περίπλοκου κειμένου που από τη μια σκοπό είχε να αντλήσει διδάγματα από την περίοδο τη κρίση για σκοπού δημοσιονομικού και να εντοπίσει μακροοικονομικέ ανισορροπίε ε, βλέποντα ε, τι επιπτώσει υπήρχαν και τι λύσει μπορούν να βρεθούν σε προβλήματα που δεν οφείλονταν στι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Τέλο πάντων ε, για να δούμε τι γίνεται με την ε, διαδικασία αυτή ολόκληρη και τη δευτερογενή νομοθεσία ε, που έχει παραμεριστεί, αυτό μας ανησυχεί. Και επίσης τα μέτρα της ανάπτυξης που έχει ορίσει ο στόχο η Προεδρία σας. Τα μέτρα για την εσωτερική αγορά. Βλέπουμε την ε, διάρθρωση της συνθήκης και εκεί δεν υπάρχει αρκετή ισορροπία. Ακόμη και αν έχουμε ως πρωταρχική μέρημνα την πειθαρχία με την έκθεση της κυρίας Φεραίρα και άλλων συναδέλφων του κυρίου Φέιο που είναι εδώ. Πρέπει να βρούμε περιθώριο και για την πειθαρχία και για άλλα πράγματα. Δεν λέμε εδώ ότι θέλουμε να γίνει ή το ένα ή το άλλο, ή η πειθαρχία ή η ανάπτυξη. Και τα δυο τα θέλουμε. Και θέλουμε μια ισορροπημένη πολιτική δημοσιονομική. Και όταν τελικά καταλήγουμε σε ένα κείμενο που δεν είναι καθόλου ισόρροπο, από οικονομική άποψη μάλλον θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβέ. Και όπω εσεί είπατε, πολλέ οικονομίε παγκοσμίω δείχνουν στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Οικονομία πόσο μερικώ υλοποιούνται ορισμένα μέτρα. Και τι θα κάνουμε τέλο πάντων, αυτό θα το, θα το κάνουμε κανόνα και με μία συνθήκη. Είναι τρέλα, καθαρή τρέλα. Και να μην σκεφτόμαστε μόνο ότι οι πιο φιλευρωπαϊστές ε, βουλευτές από το Κοινοβούλιο θα σας βοηθήσουν να περάσετε το κείμενο αυτό στα κράτη-μέλη. Είναι τρεις αυτοί που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα. Αλλά να είμαστε επικοδομητικοί εδώ. Υπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνούμε, αλλά το κείμενο δεν είναι πλήρε. Και δεν θα περάσει με τίποτα. Μια συζήτηση επί τη συνθήκη αυτή, ε, όπω είναι σήμερα, με την άποψη τη κοινή γνώμη και των κρατών μελών, δεν περνάει με τίποτα. Ακόμη και πιο φιλευρωπαϊστέ από όλου του βουλευτέ μα δεν θα μπορέσουν με τίποτα να σα βοηθήσουν. Φιλική λοιπόν συμβουλή, καθόλου απειλή, μην το πάρετε έτσι, δεν μπορεί να γίνει με βάση αυτό το κείμενο. Και μια τελευταία παρατήρηση, αν επιτρέπετε. Πέρυσι ακούσαμε και το είχα βάλει εγώ και στην εκθεσή μου τον Δεκέμβριο του 2010 ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη. Μετά μα είπαν δεν αναθεωρείται συνθήκη. Ωραία, πολύ καλά. Πολιτική επιλογή με κάποιου κινδύνου. Ε, Δευτερογενή νομοθεσία λοιπόν. Αλλά με το που τελειώνει η διαδικασία τη δευτερογενού ε, νομοθεσία, λέμε θα αλλάξουμε τη συνθήκη. Ε, μα κοιτάξτε λοιπόν, στο κοινοβούλιο αυτό ουσιαστικά μα πουλάτε εδώ και αυτή την αντίποση μα δίνετε. Δεν είναι πολύ φιλικό αυτό απέναντί μα. Εδώ έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν το λέω για σα προσωπικά, αλλά έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Να πω απλώς και εμείς τον Ιούνιο του 2010 είμαστε υπέρ της αναθεώρησης της συνθήκης και το είχαμε πει. Βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια μοίρα με εσάς. Και ακριβώ και εμά μα πούλησαν, όπω λέτε, όπω και εσά. Μα κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, πολύ εύκολο να απαντάτε έτσι, αλλά. Ακούστε με, κύριε Υπουργέ, έχετε Δέκα μέρε ακόμα. Δέκα μέρε να το πείτε ω πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ε, οι βουλευτέ να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Πείτε το. Πείτε το δυνατά και υψώστε τη φωνή σα. Εδώ ουσιαστικά θα κάνετε με μια μεγάλη χάρη σε όλη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργός. Εσείς μιλήσατε για κοροϊδία και για ξεπούλημα. Τέλος πάντων, ορισμένες χώρες που τις σχολιάσαμε και προηγουμένως, αυτές που τρόπον τεινά καθορίζουν το τι θα συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελαν μια αλλαγή στη συνθήκη και δεν πέτυχαν Τη Γερμανία εννοώ, την Πολωνία και μερικές άλλες χώρες. Ήθελαν αλλαγές στη συνθήκη. Δεν το πέτυχαν. Οπότε νομίζω λογικό είναι σε μια ένωση 27 κρατών και με τρία θεσμικά όργανα να μην κερδίζει κανείς αυτό που θέλει πάντοτε. Δεν μπορεί να κερδίζονται όλες οι μάχες. Ειλικρινώς όμως, για μας Είναι αυτονόητο ότι πάντοτε δεν θα πετυχαίνουμε. Αλλά το είχα πει και προηγουμένω για μια άλλη περίπτωση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Α είμαστε έστω ευχαριστημένοι που επιτελείται κάποια πρόοδος όσο για την ε, ανησυχία σας ότι η συνθήκη δεν είναι ισόρροπη το σχολίασα αυτό μίλησα για κάποιες προτάσεις. Προτάσεις της Πολωνίας για τη συνθήκη. Θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Σε ευχαριστώ, Σάρον. Είναι και Χριστούγεννα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω θα υπάρξουν τρει εκπρόσωποι, όλοι οι μεγάλης ε, ποιότητας, ο κ. Γκουαλτιέρη, ο κ. Περχόφτα και ο κ. Μπροκ. Ε, εάν θέλουμε να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων και αν θέλετε να ενθαρρύνετε τον Πολωνό εκπρόσωπο σε αυτέ τι συζητήσει. Για τη Γερμανία, να σα το πω αν με επιτρέπετε, ε, αισθάνομαι πολύ κοντά στη χώρα αυτή. Δεν πρέπει να δίνουμε διαρκώ την εντύπωση ότι υπάρχουν 82 εκατομμύρια Γερμανοί που είναι όλοι τη ίδια άποψη. Είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα, στην οποία και εκεί υπάρχουν εντατικέ συζητήσει. Μπορεί και εκεί να μεταβληθούν οι στάσει των μεν και των δε. Δεν μπορούμε να λέμε διαρκώ η Γερμανία. Έχω πάει μάλιστα πολλέ φορέ επίσκεψη, έχω δώσει τη δική μου μικρή συνεισφορά. Δεν μπορούμε συνεχώ να του ε, κατηγορούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τάση να λέμε ότι οι Γερμανοί έχουν διαρκώ άδικο. Όταν κάνουν κάτι δεν είναι καλό. Μόλι δεν κάνουν τίποτα πάλι έχουν άδικο. Εδώ πρέπει να επηρεάσουμε ίσω τη συζήτηση στη Γερμανία που και εντατική είναι και πιο προχωρημένη από ό,τι σε εμά, ώστε να αλλάξει η στάση που μέχρι τώρα ήταν πολύ φιλευρωπαϊκή. Δεν έχω καμία ανησυχία για τη Γερμανία προσωπικά σε ό,τι με αφορά θα εκφραστικά άσχημα. Είπα ότι η Γερμανία, όπως και η Πολωνία, όπως και το Κοινοβούλιο, θέλανε μια αλλαγή των συνδικών ήδη από τον Ιούνιο του 2010. Δεν επέκρινα λοιπόν τη Γερμανία, αντίθετα, για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο της, ε, α, της αλλαγής των συνδικών ήμουνα σύμφωνος μαζί τους. Ωραία. Ο Ούντο. Ευχαριστώ πολύ. Σάρον. Εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή αυτή, κύριε Ροστόφσκι, είναι δύο πράγματα τα οποία θυμάμαι από την Πολυλονική Προεδρία. Νομίζω είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να θυμηθεί κανείς άμα κάνει ένα δρόμο στο εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας. Καταρχήν, ήταν εκπληκτικό το βήμα προς τα εμπρός το οποίο έγινε από την Πολωνική Προεδρία ήταν η δική σας προσωπική δέσμευση ως Πρόεδρου του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια υπεράσπισης της Ευρωζώνης χωρίς καν να είσαστε μέλος της Ευρωζώνης μια εντυπωσιακή προσπάθεια να φέρετε τη χώρα σας σε μια ευρωπαϊστική θέση που πολλοί από εμά δεν την ανέμεναν καθόλου προηγουμένω. Επομένω. αυτό είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω και ως Γερμανός, ως Γερμανός σοσιαλιστής, θέλω να προσθέσω φυσιολογικά χρησιμοποιώ την μυθική μου γλώσσα αλλά τώρα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια γλώσσα η οποία είναι άμεσα κατανοητή από τους συνομιλητή μου, δεν το κάνω αυτό πολύ συχνά στην Επιτροπή μας. Συγγνώμη, <laughs> λοιπόν, Φέρνερ που μιλάω αγγλικά. Ναι, σαν Γερμανός σοσιαλιστής και Γερμανός βουλευτής θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δρόμο αυτό που ακολουθήσατε. Να μπείτε όλο, όλο και πιο βαθιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει η Πολωνία ένα μέλος της Ευρωζώνης, ελπίζω το γρηγορότερο δυνατό και σας εύχομαι να είστε πάντα από αυτούς που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η εμπειρία μου η προσωπική ήταν κάθε φορά που μιλούσαμε, κάθε φορά που ήσασταν ενώπιον αυτής της Επιτροπής ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε εσά για το μέλλον της Ευρώπης. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω δεν είναι ίσως τόσο θετικό. Αν ανατρέξω σε αυτά τα οποία συνέβαλαν οι στα οποία συνέβαλαν οι ηγέτες μας για την αντιμετώπιση της κρίσης και αυτά που έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών μας για την επίλυση της κρίσης, έχω πραγματικά σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του. Αναφέρθηκε αυτό ήδη, αλλά έχω μεγάλες αμφιβολίες για το ότι η πολιτική αυτής της αλλαγής στη συνθήκη, περιορισμένες αλλαγές που έχουν απλώς να κάνουν με την αυστηροποίηση των στοιχείων του Six Pack χωρίς όμως καμία άποψη σε αυτό το οποίο είπε ο Μάριο Ντράγκη χθες προηγουμένως ότι πρέπει να αναχαιτήσουμε το σοβαρό κίνδυνο της ύφεσης σε σχέση επίσης να βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας ώστε να βγούμε όλοι με μεγένθηση οικονομική από αυτή την κρίση, με αλληλεγγύη και με μια θετική διαδικασία επένδυσης στο ευρωπαϊκό μέλλον. Για όλα αυτά τα θέματα λοιπόν υπήρξε μηδενικό μήνυμα από το ΕΚΟΦΗΝ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σιγεία σειρμάτου και φοβάμαι ότι πολύ σύντομα οι αγορές μας την έχουν στημένη για το γεγονός αυτό ότι δεν υπήρξε κανένα μήνυμα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά του νομίσματος. Αναγνωρίζω ότι εσείς προσωπικά και η ομάδα σας, <clears throat> οι συνεργάτες σας, κάναν μεγάλες προσπάθειες για να υπερασπιστούν την Ευρώπη σε αυτή τη δύσκολη κρίση, αλλά έχω να κάνω και αυτό το αρνητικό σχόλιο, την αρνητική σύνοψη του εξαμήνου, Πρέπει να πω ότι αυτά τα οποία έκανε το Συμβούλιο σαν σύνολο για να επιλύσει την κρίση στην Ευρώπη δεν ήταν επαρκή και φαίνεται ότι θα μας φέρει μέσα σε μια πολύ δύσκολη θέση πολύ σύντομα τον επόμενο χρόνο και ελπίζω θα είσαστε από την πλευρά των Ευρωπαϊστών και θα μπορούμε να σας ε, να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσά, ακόμα και αν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ατυπικά μέτρα και να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Είναι επικίνδυνο να λέμε στα μέλη ότι έχουν χρόνο για να μιλήσουν. Θέλετε να, κάνετε μια, να δώσετε μια σύντομη απάντηση στον Ούντο. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας, τα θερμά σας λόγια. Ελπίζω ότι η Πολωνία θα είναι πάντα με τη μεριά των Ευρωπαϊστών. Δεν μπορώ να φανταστώ το αντίθετο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, <laughs> εμείς θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχει υπάρξει η επισκευή της Ευρωζώνης πρωτού μπούμε εκεί μέσα. Το βασικό όμως πρόβλημα που αναφέρατε συνδέεται με αυτό ακριβώ το ερώτημα. Όταν έχουμε μια κατάσταση στην οποία 17 χώρες σκέφτονται μονάχα το ατομικό για αυτές κόστος μιας κοινή πολιτικής, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε <clears throat> προς την κατεύθυνση της πολιτικής που θα θέλατε εσείς να δείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι το θεμελιώδες διαρθρωτικό πρόβλημα, δομικό πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό εμείς ως Πολωνία υποστηρίζουμε στεναρά περαιτέρω ολοκλήρωση, ώστε να μην λένε όλοι πάντα τι θα κοστίσει σε εμά, χωρίς να σκέφτονται τι θα τους κοστίσει η έλλειψη ή η αποτυχία δράσης ή ποια θα είναι τα ωφέλη τα οποία θα προσποριστούμε όλοι από κοινού και ο καθένας ατομικά. Τα είδαμε αυτά λοιπόν στην Πολωνία μέσα στα πλαίσια <clears throat> της διαδικασίας συνεισφοράς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν πρόσωπο με πρόσωπο όλα αυτά τα θέματα. Το ερώτημα γιατί μια μικρή, μια φτωχή χώρα όπως η, Πολωνία θα πρέπει να συμβάλλει για να υποστηρίξει την Ευρωζώνη όταν όλοι οι άλλοι είναι πολύ πιο πλούσιοι. Η απάντηση είναι απλή γιατί θα γίνουμε ακόμα φτωχότεροι αν δεν συμβάλλουμε και εμείς αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σουάμπ, πολύ θέλεις και εσύ να πεις κάτι. Τελευταία ερώτηση λοιπόν από την Ελίζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μια ακόμη φορά θέλω να συγκεντρώσω το ερώτημά μου εμπρός θέματο. Συνεχώς αναφερόμαστε στην ανάγκη ή μια ανάγκη να αλλάξει συνθήκη. Το πρόβλημα δεν θα την αλλάξουμε ή όχι, αλλά ποια είναι η ουσία της αλλαγή. Και εδώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ούντο και η Σιλβί Γκουλάρ προηγουμένως. Στο Κοινοβούλιο, όταν συζητήσαμε το Six Εργαστήκαμε επί ουσιαστικών θεμάτων και θέλουμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αν τώρα μπούμε στη δικασία αλλαγή τη συνθήκη, ότι θα περάσουν τα σωστά μηνύματα. Αναφερθήκατε σε τύχη προστασία και την ανάγκη ύπαρξή του. Στο προηγούμενό μου ερώτημα προσπάθησα να μάθω λεπτομέρειε αυτού του είδου τα τείχη. Ένα από τα τείχη προστασία που χρειαζόμαστε σχετίζεται και με τις ανισορροπίες της λειτουργίας νομισματικού τομέα και τι ανισορροπίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία 13 χρόνια. Έχουμε ανισόρροπη ανάπτυξη και ανεπαρκή γενική ανάπτυξη. Και αυτό κρύβεται σαν αίτιο, ένα από τα βασικά αίτια της κρίσης από την οποία δεν βγήκαμε ακόμα. Το θέμα της ανάπτυξης, πώς να χειριστούμε την ανάπτυξη, το κοινό νόμισμα και τη σύγκληση και το κοινό νόμισμα αυτό είναι το θέμα που ουσιαστικά θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στην αλλαγή της συνθήκης μαζί με τα άλλα τυχή προστασία. Να αντιμετωπιστούν με αλληλεγγύη τα θέματα. Αυτό δεν το βλέπουμε στις προτάσεις που υποβάλλονται από το Συμβούλιο. Και γι' αυτό ανησυχούμε τα μάλα. Εργαζόμαστε σε ένα αποσπασματικό σύμπαν. Δεν μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας και από αυτά που κάνουν άλλοι. Εδώ είναι το κομβικό σημείο για μας. Και αυτό ίσως μας οδηγήσει σε υποστήριξη ή μη υποστήριξη της αλλαγής συνθήκης. Αν η αλλαγή της συνθήκης πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, τότε εντάξει. Περισσότερο δήλωση είναι αυτό, λέει η Πρόεδρος. Ο υπουργό δεν έχει κάποια απάντηση. Είμαι Ευρωβουλευτήνα και απευθυνόμουν προ την Προεδρία. Ευχαριστώ, λέει ο Προεδρεύων. Της Εκοφή, ευχαριστώ την δήλωσή σα, Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστώ όλου. Όπω βλέπετε ε, υπάρχει πάθο όσον αφορά τη συζήτηση του θέματο τη διακυβέρνηση και τη συνθήκη. Έχουμε κοινή συζήτηση με την Επιτροπή ΑΦΚΟ αφού τελειώσουμε τι συνεδρίε τη Επιτροπής μας σήμερα το απόγευμα και εκεί θα μπούμε στο ψητό. Τι θέλει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την αλλαγή το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ που μας ξαναμιλήσατε. Σας ευχαριστώ για όλα σα κάνατε ως Προεδρία. Θα τα πούμε το απόγευμα.